Αγαπητοί συνάδελφοι, μπορούμε να αρχίσουμε γιατί ήδη έχουμε καθυστερήσει. Παρακαλώ, καθίστε για να αρχίσουμε. Έληξε η συνάντηση των συντονιστών με την συνήθη καθυστέρηση όπου αποφασίστηκε μεταξύ άλλων σας παρακαλώ συνάδελφοι, αποφασίσαμε στην Επιτροπή να ξαναδούμε τις αναφορές που σχετίζονται με το Λέιντε Κώστας, όπου ζητήσαμε τη γνωμοδότηση της ε, νομικής υπηρεσίας. Και έτσι θα εξετάσουμε το θέμα για να δούμε κατά πόσο χρειάζεται να ζητήσουμε και γνωμοδότηση άλλων επιτροπών ε, που θα αποφανθούν επί της ουσίας. Επίσης έγινε μια πρώτη συζήτηση για την ανάθεση ορισμένων εκθέσεων που ανέλαβε η Επιτροπή μας αλλά θα αποφασίσουμε στην προσεχή συνάντηση των συντονιστών. Και για την ανάθεση αυτών των εκθέσεων και για την ανάθεση ορισμένων εκθέσεων θα εφαρμόσουμε τη μέθοδο DONT. αποφασίσαμε ομόφωνα να αναθέσουμε την υπόθεση 473 κάθετος 08, την αναφορά αυτή, Klein, Atmed και θα ε, ακολουθήσουμε την οδό, τη συνήθεια οδό. Επίσης, ως προς μία πρόταση στην Ολομέλεια για την Συμφωνία Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ είπαμε ότι το θέμα αυτό θα το δούμε κατά την προσεχή συνεδρίαση και τέλος κάναμε μία αλλαγή στην ημερήσια διάταξη που θα ισχύει από την προσεχή μας συνεδρίαση, δηλαδή οι συντονιστές να συνεδριάσουν στο τέλος της πρώτης ημέρας εργασιών και όχι στην αρχή της δεύτερης. Για να μην επιβαρύνουμε κανέναν σε περίπτωση παράτασης των εργασιών. Ας περάσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης. Εάν δεν υπάρχουν άλλες παρεμβάσεις, Θα ήθελα να χαιρετήσω τις ρουμανικές αρχές που είναι παρούσες, καθώς και τους ρουμάνους πολίτες. Θα ήθελα λοιπόν να ασχοληθούμε με τις αναφορές του 17, 733 και 735 του 10 που θα δούμε από κοινού και δίνω το λόγο στον αναφέροντα, τον Κρίστη Γκόντινακ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω εκ μέρους ε, της Δημοκρατικής Συνομοσπονδίας ε, Συνδικάτων Ρουμανίας, ε, CSDR και της Ρουμανική Ομοσπονδίας Media Sint, διότι δεχθήκατε τις δύο αυτές αναφορές. Αυτό είναι σημαντικό για όλα τα μέσα ενημέρωσης στον κόσμο. Η ψηφοφορία, η απόφαση που θα λάβετε σχετικά με το θέμα αυτό θα είναι ουσιαστικής σημασίας και θα σώσει χωρίς να υπερβάλλω την δημοκρατία στην Ρουμανία. Θα ήθελα να σας παρουσιάσω την εντολή που έλαβα από τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Γιάν Μπάτσου, εξ ονόματος αυτής της Συνομοσπονδίας και των 600.000 μελών αυτής της Συνομοσπονδίας και εκ μέρους των 9.000 ε, μέλων, ε, μελών της Ρουμανικής Ομοσπονδίας Δημοσιογράφων Media Sint που μου ζητούν να μην δημιουργηθεί κυρίως ένα προηγούμενο να μην ε, θεωρούνται τρομοκράτες ε, εφεξής ε, οι Ρουμάνοι δημοσιογράφοι, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία για την, το κείμενο αυτό της 23ης Ιουνίου 2010 στο Ανώτατο Συμβούλιο της Ρουμανίας για την Εθνική Άμυνα. Θα αναφέρω αυτήν την εθνική στρατηγική εθνικής άμυνας για να μην μας κατηγορούν πλέον ότι δεν ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Παράγραφος 10 του άρθρου 6.2, ευάλωτα σημεία του κράτους. Τα, οι εκστρατείες στον τύπο που ε, κατηγορούν, επιτίθενται στα όργανα του κράτους ε, ότι, ε, ότι διαδίδουν ψευδείς πληροφορίες για να ε, για να έχουν οικονομικά ωφέλη από τα όργανα του κράτους. Όλα αυτά αποτελούν ένα στοιχείο που δημιουργεί ευάλωτα σημεία, για ευπαθή σημεία για το κράτος της Ρουμανίας. Σύμφωνα με την Συνομοσπονδία την Ευρωπαϊκή και την Διεθνή ε, των Δημοσιογράφων και των Ρεπόρτερ χωρίς σύνορα, ε, σύμφωνα με τον Νικολάη, τον Βικτόρ Μποστινά και άλλους ευρωβουλευτές και άλλα άτομα που δεν μπορώ να αναφέρω όλα εδώ, αυτή η φράση σε ένα κείμενο τόσο σημαντικό όπως την στρατηγική άμυνας μιας χώρας αποτελεί μια ε, παραβίαση της ελευθερίας έκφρασης. Οι αρχές ε, της Ρουμανίας θα διατείνονται ότι δεν ε, κατάλαβαν περί τίνος πρόκειται. Θα σας ισχυριστούν ίσως ότι δεν μπορούν να ερμηνεύσουν σωστά αυτή τη φράση. Ίσως όχι μόνο στη Ρουμανία, αλλά και σε όλες τις χώρες του κόσμου οι εκστρατείες του τύπου γίνονται κατόπιν παραγγελίας, εντολής ενός οργάνου, παραδείγματος χάρη εκστρατείες κατά του καπνού, κατά της φτώχειας, τότε οι αρχές, η κυβέρνηση, η Προεδρία, το Κοινοβούλιο μπορούν να κατακριθούν στα πλαίσια μιας τέτοιας εκστρατείας και συνεπώς δεν είναι δίκαιο να μην έχουμε πλέον το δικαίωμα να κατακρίνουμε, να μας μεταχειρίζονται όσα να είμαστε τρομοκράτες. Χρησιμοποιώ αυτή την δυνατή λέξη για έναν απλό λόγο. Διότι ε, η εθνική ασφάλεια, η παραβίαση της εθνικής ασφάλειας προβλέπει κυρώσεις δραστικές κατά των ε, δημοσιογράφων που μπορούν να καταδικαστούν σε πέντε χρόνια φυλάκιση, ε, να παρακολουθούνται να παρακολουθούνται οι τηλεφωνικές τους ε, συνομιλίες και τότε ανοίγει κανείς ε, την πόρτα σε μεγάλες καταχρήσεις. Ε, γι' αυτό πρόκειται για μεγάλη απειλή για το, την ελευθερία έκφρασης. Πρόκειται για το άρθρο 11 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, το άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Διακήρυξης των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και την απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, της 7ης Δεκεμβρίου 76 που αμφισβητείται εδώ διότι πρόκειται για μια ε, δήλωση, διακήρυξη του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που θεωρεί ότι το άρθρο 10 καθιερώνει την ελευθερία του τύπου ως θεμελιώδες δικαίωμα ε, για μια δημοκρατική κοινωνία που βασίζεται στον πλουραλισμό, το άνοιγμα δεν, αφορούν, ε, δεν αναφέρονται μόνο οι γνωμοδοτήσεις, ε, οι δηλώσεις ως ακίνδυνες, αλλά επίσης ε, πρόκειται για τοποθετήσεις που μπορεί να θεωρηθούν σκανδαλώδεις για τμήματα του πληθυσμού. Γι' αυτό το άρθρο 10 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο της Συνθήκης για την Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν παραβιαστεί. Συμπερασματικά, και εγκατακλείδη, σας παρακαλούμε να μην δημιουργήσετε εδώ ένα προηγούμενο με την περίπτωση της Ρουμανίας. Εμείς ως αναφέροντες δεν θέλουμε ε, να τιμωρηθεί το κράτος, να επιβληθούν κυρώσεις στο κράτος, διότι εμείς πληρώνουμε, καταβάλουμε μια, ε, ένα πρόστιμο. Ε, έχουμε τιμωρηθεί εδώ με αυτό, αλλά θέλουμε να σταλεί ένα μήνυμα στις αρχές της Ρουμανίας, ούτω ώστε από τη στρατηγική εθνική Άμυνα να αφαιρέσουν αυτή τη διάταξη που είναι επικίνδυνη για την ελευθερία έκφρασης. Διότι έχουμε άλλα πράγματα να κάνουμε. Πρέπει να αποπολιτικοποιήσουμε τα δύο όργανα ε, της δημόσιας τηλεόρασης και του δημόσιου ραδιοφώνου να μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη προστασία, μια πραγματική προστασία για τους δημοσιογράφους και όχι όπως συνέβη πριν μερικές μέρες στον τοπικό τύπο. Ο επικεφαλής της εργοδοσίας του ρουμανικού τύπου κατηγορήθηκε. Υπάρχουν πάρα πολλές καταχρήσεις ε, κατά των δημοσιογράφων στη Ρουμανία και μαζί μπορούμε να βρούμε μια λύση για να τους βοηθήσουμε. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και δίνω τον λόγο ε, στην συνάδελφο από την Συνομοσπονδία των ε, Δημοσιογράφων. Ναι, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η ε, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων αντιπροσωπεύει τους δημοσιογράφους όλης της Ευρώπης και είμαι εδώ για να υποστηρίξω αυτήν την αναφορά διότι πρόκειται για μια ευκαιρία που έχει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασχοληθεί με την προάσπιση της ελευθερίας του τύπου στην Ευρώπη κυρίως στα νέα κράτη-μέλη. Γιατί Έχουμε αυτήν την συγκεκριμένη περίπτωση που μας ανησυχεί διότι λέγοντας ότι το κράτος είναι βάλωτο απέναντι στους δημοσιογράφους ε, θέλουν να σιωπήσουν οι ε, δημοσιογράφοι να εφαρμόσουν την αυτολογοκρισία που είναι ένα δηλητήριο στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επιδιώκουν να ανατρέψουν μια κατάσταση νομική, να ανατρέψουν το τεκμήριο της απόδειξης. Ποιος είναι βάλωτο οι δημοσιογράφοι ή οι πολιτικοί, ποιος αναλαμβάνει τον κίνδυνο για να πληροφορεί, να ενημερώνει ημερών. Λοιπόν, οι δημοσιογράφοι ή οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε σαφείς, να έχουμε έναν νόμο ε, που, την, ε, που να ε, προσωμιάζει το αδίκημα της γνώμης με το αδίκημα της τρομοκρατίας. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό. Αυτό προκαλεί ε, μίσος, ε, μίσος ε, ρατσιστικό και γι' αυτό ελπίζουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει τις αναφορές αυτές και ότι θα τις παρεπέμψει βάση στο άρθρο 11 της Χάρτας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων που περιλαμβάνει την ελευθερία του τύπου όχι μόνο προς όφελος των Ρουμάνων πολιτών και των Ρουμάνων δημοσιογράφων, αλλά προ όφελο και των άλλων κρατών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, εφόσον η Ρουμανία δεν είναι δυστυχώ η μόνη χώρα όπου ασκούνται πιέσει εμπορικέ και πολιτικέ πάνω στους δημοσιογράφους ενώ ε, το απόρριτο της πηγής ε, απειλείται και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να ασχοληθείτε με το πρόβλημα αυτό το συντομότερο δυνατόν, δηλαδή τώρα. Ε, εν κατακλείδη η Ομοσπονδία μας θα εξετάσει εντελεχώς την κατάσταση των δημοσιογράφων στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στην Ρουμανία και αυτό θα γίνει ε, συγκεκριμένα τον Ιανουάριο 2011 με το Συνδικάτο MediaSint στην Ρουμανία. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ και δίνω το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επίτροπης. Ροντρίγκο Μπαλεστέρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η Επιτροπή έχει, πλή, έχει συνειδητοποιήσει την κατάσταση αυτή και την μεγάλη ανησυχία που δημιούργησε στην Ρουμανία όπου μέλη της κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής τάξης ανησυχούν. Έχει δεσμευθεί η Επιτροπή να προασπίζεται την, ε, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την ελευθερία έκφρασης. Αυτό είναι σημαντικό και αυτό μπορούμε να το κάνουμε βεβαίω μόνο μέσα στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας. Σύμφωνα με το άρθρο 51 ε, του χάρτη, οι διατάξεις του χάρτη χάρτη αναφέρονται σε όργανα, σώματα ε, της Ένωσης αφενός και αφετέρου. Επίσης αφορούν τα κράτη-μέλη μόνον όταν ε, εφαρμόζουν ε, νομοθεσία κοινοτική. Σε αυτήν την περίπτωση η Ρουμανία δεν εφαρμόζει εδώ καμιά νομοθεσία κοινοτική. Συνεπώς πρέπει μόνο η Ρουμανία, να πόκειται στην Ρουμανία να εκπληρώσει τις ε, υποχρεώσεις σχετικά με την ελευθερία ε, έκφρασης που απορρέουν από διεθνή ε, υποχρεώσεις, συμβατικές υποχρεώσεις. Ο πλουραλισμός των μέσων και η ελευθερία του τύπου αποτελεί ένας από τους πυλώνες της δημοκρατικής κοινωνίας. Ο πλουραλισμός, η προστασία των δημοσιογράφων, προστασία των πηγών ε, των δημοσιογράφων, τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης ε, και τα ρυθμιστικά σώματα είναι ουσιώδη στοιχεία για την ελευθερία της έκφρασης. Όπως η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ είχε ήδη την ευκαιρία να το πει σε αυτήν την Επιτροπή, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης είναι μια ευκαιρία για την Ευρώπη και δεν είναι απειλή για την εθνική ασφάλεια. Ευχαριστώ πολύ. Ένα λεπτό κύριε Μποστινάρο. Δίνω το λόγο στο Βαλέριο Τούρκαν που εκπροσωπεί την κυβέρνηση. Κύριε Κυρία Πρόεδρε, αξιότιμες κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, θα ήθελα πρώτα να ευχαριστήσω όλους και όλες τις Ευρωβουλευτές μέλη της Επιτροπής Αναφορών για την ευκαιρία που προσφέρουν στις ρουμανικές αρχές να διευκρινίσουν το θέμα. Αντιμετωπίζεται δύο αναφορές που περιέχουν παραπλανητικές πληροφορίες. Είμαι πρώην δημοσιογράφος και σήμερα βέβαια εκπροσωπώ τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Μαζί μου ο κύριος Μπογκδάν Μανόγιου, Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Οι αναφορές δεν έχουν αυστηρό περιεχόμενο και δεν αποπνέουν σωστά το πνεύμα των ε, κειμένων στα οποία παραπέμπουν. Ε, θα συνεχίσω όμως στη ρουμανική γλώσσα, αν μου επιτρέπετε. Αγαπητές κυρίες και κύριοι ευρωβουλευτές, η εθνική στρατηγική η άμυνας δεν λέει πουθενά ότι μπορούν να οδηγήσουν σε τροτότητα της εθνικής άμυνας τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Πρόκειται ωστόσο για παραπλάνηση, για παραπλάνηση των Ευρωβουλευτών. Η στρατηγική της Εθνικής Άμυνας δεν αναφέρεται παρά μόνο σε εκστρατείε τύπου οι οποίε είναι βασισμένε σε παραπληροφόρηση και έχουν ως στόχο να δυσφημίσουν τις εθνικές αρχές θέτοντα σε κίνδυνο έτσι και, το, και την εικόνα και τι δραστηριότητε των δημοσίων αρχών. Δεν αναφερόμαστε στα μέσα στο σύνολό τους. Τι βλέπουμε στο κείμενο. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα από μια πλευρά στην κατάσταση των αναφερομένων και στα κείμενα, στα πρωτότυπα κείμενα. Οι αναφερόμενοι έχουν περιλάβει μέσα στα, στις αναφορές τους ορισμένες παραθέσεις σε εισαγωγικά χωρίς να εξηγούν από πού τις πήραν. Λέγουν ότι τα μέσα οδηγούν ε, σε τροτότητα των ρουμανικών δημοσίων αρχών. Πρόκειται για παραβίαση των κανόνων διοντολογίας του δημοσιογραφικού επαγγέλματος. Πώς είναι δυνατόν αυτό να θεωρηθεί νόμιμο σε οποιαδήποτε χώρα μέλος. Ένας μεγάλος αριθμός επαγγελματικών οργανώσεων και δημοσιογράφων στην Ρουμανία εξέφρασαν τις ανησυχίες τους σχετικά με τον ενδεχόμενο εκβιασμού, με μυστικές εκστρατείες που απευθύνονται στους ε, ε, θεατές, οι τηλεθεατές, οι ακροατές των ε, ρουμανικών ε, δημοσίων μέσων ενημέρωσης. Πρόκειται λοιπόν για παραπληροφόρηση. Ένας μεγάλος αριθμός των εκστατιών αυτών του τύπου ξεκινούν από πρόσωπα τα οποία προσπαθούν να αποκτήσουν οικονομικό όφελος ή που προσπαθούν να ασκήσουν πίεση σε αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις, τους νομοθέτες ή αυτούς που ασκούν την πολιτική στη Ρουμανία. Έχουμε γνωρίσει πολλέ τέτοιε περιπτώσει στη Ρουμανία. Πριν από λίγε εβδομάδε το Εθνικό, Συμβούλιο, το Εθνικό, Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο επέβαλε πρόστιμα σε δύο ε, κανάλια τηλεοπτικά και μάλιστα και σε, έναν, σε ένα από του διευθυντέ ενό τέτοιου καναλιού. Η Εθνική Άμυνα δεν επιβάλλει κανένα απολύτω περιορισμό στα μέσα μαζική ενημέρωση. Αυτή είναι η συνολική μα άποψη την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να την ερμηνεύσει κανείς ως ανάλυση ενός κινδύνου για την δημοκρατία, εφόσον αυτός ε, υπάρχει. Υπάρχει ένα παράδειγμα. Το 2009 το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο εξέδωσε δεκάδες αποφάσεις κυρώσεων κατά τηλεοπτικών καναλιών διότι δεν έδιναν το δικαίωμα απάντησης ή διότι εξέπεμπαν ε, αθεμελίωτες κατηγορίες και μάλιστα για δύο ε, τηλεοπτικά κανάλια τα οποία προβαίνουν διαρκώς και συστηματικά σε εκστρατείες δυσφήμισης. Αυτό δεν χαρακτηρίζει βέβαια όλο το ρουμανικό τύπο, ωστόσο είναι ένα φαινόμενο που λαμβάνει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια εκστατείες από, τον, από τα μέσα ενημέρωση. Το κεφάλαιο για την τροτότητα αυτή δεν αναφέρεται μονάχα στην εθνική άμυνα. Πρόκειται για μια ε, τροτότητα που έχει εντοπιστεί στο πολιτικό επίπεδο και στην ε, ρουμανική κοινωνία γενικότερα και που θίγει ολόκληρη τη Ρουμανία. Όχι μόνο για, τις, για την εθνική άμυνα Για παράδειγμα, η λειτουργία των δημοσίων αρχών, μειωμένη διοικητική ικανότητα, η ανάπτυξη των περιφερειών. Το ίδιο και για τα ίδια τα κόμματα. η ε, υπερβολική πολιτικοποίηση των θεσμών. Τέτοιες είναι οι κατηγορίες που ακούγονται από ενορχιστρωμένες εκστατείες των μέσων ενημέρωσης. Το Ρουμανικό Σύνταγμα διευκρινίζει ότι τα μέσα ενημέρωσης, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, οφείλουν να προσφέρουν αξιόπιστες πληροφορίες στο κοινό. Αυτές οι δηλώσεις που έχουν γίνει ωστόσο μέχρι τώρα σχετικά με τις δημόσιες αρχές και τις ε, ε, ένοπλες δυνάμεις δεν μπορούν να οδηγήσουν σε μια υγιή συζήτηση. Κρίσεις και επικρίσεις χωρίς καμία θεμελίωση δεν μπορούν να νομιμοποιούνται. Χρειάζεται πάντοτε να υπάρχει συγκεκριμένη θεμελίωση και η συγκεκριμένη θεμελίωση χρειάζεται επίσης και για τις αναφορές ενώπιον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Το Ρουμανικό Σύνταγμα επιτρέπει την ελευθερία έκφρασης. Ο τύπος έχει την δική του δεοντολογία. Η Εθνική Άμυνα δεν, δεν θα επιβάλλει κανένα περιορισμό στη ρουμανική δημοσιογραφία. Παρόλο που έχει την δική του διοντολογία ο τύπος, δεν εμποδίζει στο πολιτικό επίπεδο να γίνουν ορισμένες διαπιστώσεις. Υπάρχουν αρνητικά φαινόμενα και στον τύπο που καμιά φορά αναγκάζουν να γίνει μια πολιτική συζήτηση η οποία ενδεχομένως βλάπτει την δημοκρατία. δυστυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να διαπιστώσουμε ότι γίνεται απόπειρα παραπλάνησης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σας ευχαριστώ πολύ. Αρχίζει η συζήτηση. Η κυρία Άουκεν ζήτησε το λόγο. Thank you very much. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω δύο σχόλια να κάνω, αφενός προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Πώς, ε, δεν, πώς θεωρείτε ότι δεν εμπίπτουν στο κοινοτικό δικαιικό σύστημα τέτοια θέματα. Βέβαια ο χάρτης αναφέρεται μοναχά στα θεσμικά όργανα, αλλά η συνθήκη όπως είπατε και εσείς είναι τόσο σημαντική. Και εφόσον παραβιάζεται η συνθήκη, η οποία καθαρά παραβιάζεται εν προκειμένου, εμείς οφείλουμε να ασχοληθούμε με το και να εγγύψουμε στο θέμα αυτό. Και έχω την εντύπωση πραγματικά ότι υπονομεύεται τη εξουσία του Κοινοβουλίου. Αλλά ταυτόχρονα υπονομεύετε και του εαυτού σα, εσεί, η Κομισιόν δηλαδή, αρνούμενοι να, βάλε, να λάβετε υπόψη σα. Μα σοβαρά το λέω. Πολύ σοβαρά αυτέ τι κατηγορίε. Πρέπει να καταστήσουμε σαφέ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι εμεί θεωρούμε τόσο σημαντικά τα θεμελιώδη δικαιώματα για την Ευρωπαϊκή Ένωση που ασφαλώς και πρέπει να επιληφθούμε. Και τώρα θα έρθω στο δεύτερο σχόλιο. Ακούγοντα τον εκπρόσωπο τη ρουμανική κυβερνήσεω, λυπούμε πολύ που είμαι υποχρεωμένο να το πω, ήταν ε, σαφέστατο ότι κάτι, πολύ, κάτι πάει πολύ άσχημα στη ρουμανική ε, δημοκρατία. Όλε οι χώρε μέλη. Α, οι καημένοι πολιτικοί, οι καημένε οι κυβερνήσεις, οι καημένοι θεσμοί που φύγονται και πλήττονται από δημοσιογραφικέ εκστρατείες. Μακάρι να μπορούσαμε να τους κλείσουμε όλους αυτούς, αλλά δεν μπορούμε. Όλες οι αρχές ελευθεροτυπίας, ελευθερίας έκφρασης, δεν επιτρέπουν να τους κλείσουμε τα στόματα. Μπορούμε να τους αντιμετωπίσουμε με τα ίδια μέσα, αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την κρατική εξουσία για να κλείσουν αυτές τις ε, αυτά τα δημοσιογραφικά στόματα γιατί τότε πέφτουμε στη χειρότερη δικτατορία. Αυτό είναι υποχρεωμένη να πω στη ρωμανική κυβέρνηση. Και μάλιστα με πολύ εμφαντικό και αυστηρό τρόπο. Πρόκειται για ξεκάθαρη περίπτωση μιας χώρας που προσπαθεί να αρνηθεί βασικές θεμελιώδεις αρχές και ελευθερίες της Ένωσης. Το μόνο που λέτε είναι ότι έχετε απέναντί σας, αντιμετωπίζετε δηλαδή, αρνητικές διαφημιστικές εκστρατείες. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε με επιχειρήματα, αλλά ποτέ με την κρατική βία και εξουσία. Εσείς κύριε Μποστινάρου τώρα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμες αρχές της ε, ρουμανικής κυβέρνησης. Συνάδελφοι, σήμερα δεν μιλάμε για μια κατάσταση η οποία αφορά μια χώρα η οποία θα προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν μιλάμε για μια χώρα της Ανατολής, της Λατινικής Αμερικής, δεν μιλάμε για τη Ρωσία ή την Κίνα. Μιλάμε για μια χώρα που είναι πλήρες μέλος από την 1η του 2007 που στη συνθήκη της Κοπενχάγης η ελευθερία τύπου και η ελευθερία των ΜΜΕ ήταν πρόκριμα για να μπορέσει κανείς να προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στα πλαίσια της υπεράσπισης του τύπου και αν δεν υπήρχε αυτή, αν δεν γινόταν αυτή η υπεράσπιση τότε κανείς δεν θα μπορούσε να προσχωρήσει μετά 21 χρόνια μετά τη Ρουμανική Επανάσταση θα πρέπει πάλι να προασπιζόμαστε την ελευθεροτυπία που θα έπρεπε να είναι ένα αυτονόητο αγαθό. Οι αναφέροντες δεν σχετίζονται με μία ομάδα ε, δημοσιογράφων της ε, Ρουμανίας όπως προσπαθεί να προωθήσει η κυβέρνηση. Μιλάμε για την τήρηση της χάρτας των θεμελιωδών δικαιωμάτων όπως επικυρώθηκε από τη ρουμανική κυβέρνηση. Επιπλέον, οι δημοσιογράφοι χωρίς σύνορα όρισαν παραβιάσεις στην ελευθεροτυπία της Ρουμανίας μέσα στα πλαίσια αυτού του εθνικού νόμου. Επίσης, το Ανώτατο Συμβούλιο, το Συμβούλιο Επικρατείας ασχολήθηκε με αυτό το θέμα και όρισε ότι πρόκειται για δραστηριότητες εκφοβισμού. Αλλά δυστυχώς το κράτος δεν κινητοποίησε όλες τις θεσμικές αρχές για να συζητήσει αυτό το θέμα της ελευθεροτυπίας. Αναφερθήκατε στο άρθρο 6 παράγραφος 2. Θα ήθελα να σας ε, υπενθυμίσω και να υπενθυμίσω στη ρουμανική κυβέρνηση ότι καμία χώρα δεν έχει έναν τέτοιο παράλογο νόμο η κοινοπολιτεία των ανεξαρτήτων κρατών της ε, Ρωσίας δεν έχει έναν τέτοιο απαράδεκτο νόμο. Πώς μπορεί να τον έχει μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, λέγεται ότι αυτός ο νόμος είναι άκακος και ότι κανένας δεν έχει πληγή από αυτό. Όμως, ο Τεοντόρ Στολοζάν μας είπε ποιος είναι ο στόχος αυτής της δράσης και αναφέρομαι στο έγγραφο το οποίο διαβίβασε ο πρόσωπος του ΠΕΛΤΕ στη Ρουμανία. Υπάρχουν η ρεαλιτάτεα και η αντένα τρέι οι οποίες λειτουργούν και δυστυχώς μεροληπτούν για να διασύρουν την κυβέρνηση και ιδιαίτερα τον πρόεδρο Μπασέσκου. Εδώ είναι το πρόβλημα. Δηλαδή γίνεται λόγος για τη στάση ορισμένων δημοσιογράφων. Δεν μπορεί κανείς να κατακρίνει την κυβέρνηση. αυτή η, αυτός ο νόμος δεν μιλάει για στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα, για απόρριτα στοιχεία, για πώληση μυστικών του ε, αμυντικού συμφώνου, για τρομοκρατία κατά του ΝΑΤΟ, ας πούμε. Απλώς ε, γίνεται λόγος για ευαλωτότητα του κράτους και μεροληψία των δύο καναλιών. Και αυτό μας λέει και ο Στολοζάν, ότι δεν του αρέσει η στάση των δημοσιογράφων. Θα ήθελα να ρωτήσω τον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εάν δεν θα έπρεπε να τα γνωρίζει όλα αυτά. Και μην ξεχνάτε τι είπε και η κυρία Ρέντινγκ. Η κυρία Βίβιαν Ρέντινγκ, αντιπρόεδρος Επιτροπής, είχε πει όταν ρωτήθηκε για τον τύπο της ε, Ρουμανίας με ανησυχή κατάσταση στη Ρουμανία. Όταν μία αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής λέει ότι ανησυχεί για την κατάσταση μιας χώρας, δεν είναι απλώς ανήσυχη χωρίς να υπάρχει τίποτα, χωρίς να υπάρχει ουσία. Λαμβάνει υπόψη τις καταχρήσεις που έχουν γίνει και τον παραλογισμό. Πρόκειται για μία προκατάληψη, διότι εμείς έχουμε επισύρει την προσοχή σας σε αυτό το θέμα και σας λέμε ότι, θα πρέπει να αφαιρεθεί αυτή η παράγραφος από την ε, συμφωνία από τον νόμο αυτό αμυντικής στρατηγικής. Ο Σούλτς, ο Βότσον και η Κον απέστειλαν μία επιστολή προς τη ρουμανική κυβέρνηση ζητώντας να αποσυρθεί αυτή η παράγραφος. Ούτε καν ελήφθη υπόψη αυτή η θέση. Δεν μιλάμε λοιπόν για κυρώσει. Δεν πρέπει να ε, πληρώσει η ρουμανική κυβέρνηση. Απλώς θα πρέπει το ρουμανικό κοινοβούλιο να αποσύρει αυτό το άρθρο. Γιατί Μόνο έτσι θα επανέλθει η τάξη και θα μπορέσουμε να συμβαδίζουμε με την κοινοτική ένωμη τάξη. Αλλιώς καθίσταται σαφές ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν μπορεί να εθελοτυφλεί μπροστά σε αυτή την κατάσταση και θα ήθελα να παραμείνει αυτή η αναφορά ανοιχτή μέχρι ότου μάθουμε τι θα ψηφίσει το Ρουμανικό Κοινοβούλιο και μετά θα δούμε ποιες θα είναι οι μελλοντικές μας δράσεις. Ευχαριστώ. Κολέγα Μέγερ. Μέγερ, ευχαριστώ. Θα ήθελα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου προς τους αναφέροντες, διότι έχουμε να κάνουμε με κάτι το πολύ σοβαρό. Εγώ κατανόησα απόλυτα την παρέμβαση της Ρουμανικής κυβέρνησης και νομίζω ότι και η ερμηνεία της κυβέρνησης είναι πολύ σοβαρή, διότι δεν ξέρω καμία χώρα από τις 27 όπου η εκτελεστική ε, εξουσία δεν επιτρέπει την ελεύθερη επικοινωνία. Στη Ισπανία κάτι τέτοιο το αναλαμβάνει η δικαστική εξουσία. Δηλαδή το εκτελεστικό δεν μπορεί να είναι και δικαστική εξουσία. Βεβαίω μπορούμε να μιλήσουμε για το πώς γίνονται τα πράγματα και τι ισχύει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω πρόβλημα. Συμφωνώ με τον κύριο Μποστινάρ. Δεν ξέρω να υπάρχει ένας τέτοιο νόμος αμυντικής στρατηγικής. Και ο νόμος αμυντικής στρατηγικής δεν ασχολείται με, με τα ΜΜΕ, στη χώρα μου τουλάχιστον. Και με όλες τις δημοσιεύσεις του Wikileaks όπου εμπλέκονται όλες οι κυβερνήσεις και η δική μου κυβέρνηση. Με αυτό το νόμο που έχετε θα έπρεπε να κλείνατε κάθε κανάλι, όλο τον τύπο, να μην υπήρχε ελευθεροτυπία, να έκλειναν όλα. Η ελευθερία επικοινωνίας και η ελευθερία ε, έκφρασης είναι θεμελιώδης ε, ανάγκη και μόνο μια δικαστική εξουσία μπορεί να αποφανθεί επί παρομοίων θεμάτων. Διότι μία εκστρατεία σπήλωσης ίσως αφορά ενημέρωση από τα ΜΜΕ για ένα θέμα το οποίο δεν αρέσει στην ρουμανική κυβέρνηση. Έχει δίκιο κυρία Άουκεν όλες οι κυβερνήσεις είναι νευρικές ως προς τα ΜΜΕ. Ποια κυβέρνηση είναι ευχαριστημένη με τα ΜΜΕ, καμία. Γιατί υφίσταται κριτική. Θα ήθελα λοιπόν η ρουμανική κυβέρνηση να λάβει υπόψη ότι αυτός ο νόμος αμυντικής στρατηγικής δεν έχει καμία σχέση με τα ΜΜΕ. Θα πρέπει να παραμείνει η αναφορά ανοιχτή, να δούμε τι θα ψηφίσει η ρουμανική κυβέρνηση, το ρουμανικό κοινοβούλιο και αν δεν υπάρξουν αυτά αποτελέσματα τότε θα εργαστούμε διαφορετικά. Δηλαδή στο Συμβούλιο θα, θα, θα ζητήσουμε το Συμβούλιο να αποφανθεί και θα ζητήσουμε να αντιδράσει και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διότι είναι ανήκουστος ένας τέτοιος νόμος φήμωσης των ΜΜΕ. Ουγγουρεάνου. Παρακαλώ πολύ, δεν θέλω χειροκροτήματα εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά είναι καλοδεχούμενη, διότι οποιαδήποτε ε, ζωντανή συζήτηση για την ε, κατάσταση του τύπου σήμερα είναι υγιής και βεβαίως άπτεται πραγματικά της ουσίας της δημοκρατίας. Είναι καλοδεχόμενη λοιπόν η ε, συζήτηση αυτή. Όπως είπε βέβαια ο διακεκριμένο εκπρόσωπο της ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν εμπίπτει σε ευρωπαϊκέ αρμοδιότητες. Νομίζω ωστόσο ότι η συζήτηση αυτή πρέπει να λάβει χώρα ανοιχτά. Νομίζω τα γεγονότα είναι σαφή και απλά. Πρώτα, δεν υπάρχει κανένας νόμος κατά της δημοσιογραφίας ή των δημοσιογράφων στη Ρουμανία. Η εθνική ασφάλεια δεν είναι νόμος, αυτό είναι γεγονό. Η εθνική ασφάλεια είναι τμήμα ενός εθνικού δόγματος που υποβλήθηκε στη Ρουμανική Βουλή, θα εγκριθεί ή θα απορριφθεί, αλλά δεν μπορεί να είναι ούτε κείμενο ούτε κώδικα νόμου. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να σας επισημάνω τώρα ποιες είναι πραγματικά οι περιστάσεις, η πραγματικότητα δηλαδή του δημοσιογραφικού κόσμου στη Ρουμανία. Μετά από το 2005 ουδής δημοσιογράφος εδιώχθη ή υπέστη δίποτε βλάβη γιατί εξέφρασε την άποψή του. Κανένας ραδιοφωνικός ή τηλεοπτικός σταθμός ή εκδοτικός οίκος εφημερίδων ούτε άλλωστε καμία ιστοσελίδα έκλεισε ή ε, απειλήθηκε με διοικητικές πράξεις. Δεν είμαστε Ρωσία όπου ε, σημειώνονται φόνοι δημοσιογράφων σχεδόν κάθε μήνα. Νομίζω ότι η Ρουμανία είναι ενδιαφέρον παράδειγμα. Δεν έχουμε πρόβλημα με την ελευθερία του τύπου. Αντιθέτως, η Ρουμανία είναι μια χώρα που ίδιος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχασε ενώπιον του δικαστηρίου αγωγή περί δυσφημίσεως κατά δημοσιογράφου. Και αυτό πάλι γεγονό είναι και είναι τμήμα της νομολογίας των ρουμανικών δικαστηρίων. Αν με επιτρέπετε να πω, η συζήτηση αυτή είναι, η δημοσιογραφία είναι καμιά φορά ε, ευφυής, αλλά πάντοτε είναι ελεύθερη. Μπορεί να τα λέει με τρόπο ε, πικάντικο, αλλά πάντως είναι, όπως είπα, είναι μια επαγγελματική δημοσιογραφία με χαρακτήρα αλλά ελεύθερη και έχει προσφέρει καλό τα τελευταίες, τελευταίες δύο δεκαετίες στη Ρουμανία. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ συνάδελφος Πρέντα. Ε, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν είμαι ιδιαίτερα ευτυχής με αυτά που είπε ο συνάδελφος, διότι Πρόκειται για μία συζήτηση που λαμβάνει η χώρα στη Ρουμανία και το θέμα έχει σχέση με μία ιδιαίτερα πολιτικοποιημένη συζήτηση στη Ρουμανία. Η ελεύθερη έκφραση είναι το διακύβευμα. Γιατί δεν μιλάμε για τον τύπο αποκλειστικά. Πρόκειται για μια πολιτική εκστρατεία πολιτικών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν ε, τον τύπο. Δηλαδή, πρόκειται για την ε, κατάσχεση των ε, δυνατοτήτων έκφρασης του τύπου. Δεν πρόκειται για μια εκστρατεία κατά του καπνού. Πρόκειται για μια εκστρατεία σπήλωσης ορισμένη πολιτικοί χρησιμοποιούν τον τύπο στη Ρουμανία για να εξαγοράσουν τη συνείδηση των ανθρώπων. Αυτή είναι η στάση ορισμένων πολιτικών. Και έτσι βλέπουν οι περισσότεροι πολιτικοί τον τύπο. Δηλαδή βλέπουν τον τύπο ως υποχείριο της θέλησή τους. Δηλαδή ταπεινώνουν τον τύπο και λένε ότι οι δημοσιογράφοι δεν ε, είναι σε θέση να εκφράσουν μία σωστή γνώμη. Αυτή είναι η στάση των πολιτικών στη Ρουμανία, οι οποίοι αγνοούν τον τύπο, εκτός και αν τον έχουν υποχείριο. Πρόκειται για την σπήλωση του τύπου από ένα μέρος ε, του πολιτικού κόσμου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πρέπει να υποστηρίξουμε αυτή την αναφορά. Είναι απαράδεκτη η κατάσταση που μας οδηγεί στο να τρέξουμε σε δικτατορικά καθεστώτα. Η κυρία Γκρουνή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Είναι περίπλοκη η συζήτηση. Δεν ζούμε στη Ρουμανία, δεν έχουμε τις αποδείξεις που θα ήταν απαραίτητες ο καθένας προβάλλει τα επιχειρήματά του, είναι λίγο δύσκολο το θέμα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην απάντησή της, όπως βέβαια ζητήσαμε μια ταχεία εξέταση, ίσως δεν είχαν και πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να εξετάσουν, να φωτίσουν από όλες τις πλευρές το θέμα. Εγώ είμαι Γαλλίδα βέβαια. Στην Γαλλία ακούω επίσης συχνά ότι φημώνεται ο τύπος από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας μας. Εγώ διαβάζω πολύ τις εφημερίδες, βλέπω την τηλεόραση. Μάλλον διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν φήμωνε ο πρόεδρος τον τύπο, αυτή τη γνώμη έχω. Δεν θέλω βέβαια να στιγματίσω την Ρουμανία. Είναι πάντα, πάντα ευαίσθητα τα θέματα αυτά και ιδιαίτερα έντονου πολιτικού χαρακτήρα. Θα προτιμούσα όπως λέω και πάντοτε, να έχουμε μια πιο αντικειμενική ματιά πάνω στην ελευθερία του τύπου και θα συμβούλευα να κάνουμε μια συζήτηση επί της ελευθερίας του τύπου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι στοχευμένα ειδικά στην Ρουμανία. Νομίζω ότι το θέμα είναι ουσιαστικό. Δεν είναι και απόλυτα διευκρινισμένο ότι εμπίπτει στις αρμοδιότητές μας αλλά είναι θέμα δημοκρατίας και νομίζω μπορούμε να το συζητήσουμε και πολύ πιο ευρέως και πιο γαλήνια. Ευχαριστώ. Ο συνάδελφος Λίκονλα. Εξ ονόματος ε, της ομάδας των φιλελευθέρων. Θα μιλήσω τώρα ρουμανικά. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να κάνω ορισμένες διευκρινήσεις νομικής υφής έτσι ώστε η Επιτροπή σας να ε, γνωρίζει την υφή και τη φύση αυτής της αναφοράς. Η Εθνική Αμυντική Στρατηγική ε, είναι ένα πολιτικό έγγραφο το οποίο προβλέπεται από το Ρουμανικό Σύνταγμα που τη στιγμή που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο έχει νομική ισχύ. Αφορά την ασφάλεια του Ρουμανικού κράτους και σχετίζεται με βασικές αρχές οι οποίες έχουν εγκριθεί στα πλαίσια της ε, ασφάλειας και της άμυνας της χώρας. Αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να προβούμε σε μία μεταρρύθμιση του πλαισίου σε σχέση με την παραβίαση του ευρωπαϊκού δικαίου. Θα ήθελα να κάνω την εξής ε, παρατήρηση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στο άρθρο 200 σε σχέση με το, το γράμμα δηλαδή του συντάγματος γίνεται λόγος για συμμετοχή στα ανθρώπινα δικαιώματα και ε, έγκριση νόμου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε κατά πόσο αυτό το, το γράμμα του νόμου παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα ως προς τις προβλέψεις της συνθήκης της Λισαβόνας θα ήθελα να αναφερθώ στο άρθρο 6, τελευταία παράγραφο, που ζητά από την Ένωση να λάβει τα κατάλληλα μέτρα για ε, τα, για την επίλυση ζητημάτων όσον αφορά την ε, τήρηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και έτσι θα πρέπει, εκεί θα πρέπει να εντάξουμε την ε, εν λόγω αναφορά. Στο άρθρο 6 της συνθήκης, σε σχέση με τις ε, κυβερνητικές δηλώσεις, δεν θα πρέπει παρά να πω το εξής. Εάν θεωρείτε ότι αυτή η εκστρατεία κατά του τύπου θέλει να οδηγήσει σε ευεργετήματα υπέν ορισμένων ανθρώπων, τότε αυτό αποτελεί ποινικό αδίκημα. Και νομίζω ότι εάν δεν υπάρχει τέτοια ε, δικαιοσύνη στη Ρουμανία, τότε θα πρέπει να την δημιουργήσουμε. Μόνο η δικαστική εξουσία μπορεί να αποφανθεί. Και νομίζω ότι αυτό που θα πρέπει να προασπίσουμε είναι θεμελιώδη δικαιώματα. Αυτό που συνέβη χτες στην Επιτροπή ήταν πολύ ε, σοβαρό. Δηλαδή αποκαλύπτηκαν έγγραφα υπομορφή στενογραφίας. Ο ρουμανικός νόμος και το ποινικό δίκαιο απαγορεύει να χρησιμοποιηθούν στοιχεία ενός φακέλου τη στιγμή που δεν έχει αποφανθεί ένα δικαστήριο. Δυστυχώς οι τηλεφωνικές υποκλοπές στη Ρουμανία είναι καθημερινή κατάσταση. Δηλαδή καθημερινά γίνονται υποκλοπές χωρίς κανένας να αναφερθεί ποτέ στην νομιμότητα αυτών των υποκλοπών που στη συνέχεια ε, χρησιμοποιούνται στους ε, δικαστικούς φακέλους. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς ε, λειτουργεί το δίκαιο σε ορισμένες χώρες. Γιατί υπάρχει πολιτική μεροληψία και ε, όχι δημοσιογραφική μεροληψία. θα πρέπει ένα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιτρέπει την ελευθερία έκφραση των ΜΜΕ. Αυτής, αυτές είναι οι ευρωπαϊκές αρχές. Και δεν θα πρέπει να υπάρχει ε, εθελοτυφλία και στρούθοκαμιλισμός όταν υπάρχει μια τέτοια στάση της, ε, του ρουμανικού πολιτικού κόσμου. Θα πρέπει ο φάκελος να παραμείνει ανοιχτός και θα πρέπει να τηρηθούν οι ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Ελπίζω εσείς να συμμερίζεστε αυτές τις αρχές όπως θέλουμε να τις ε, συμμεριστούμε κι εμείς. Hefner. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε μπροστά σε μια σοβαρή κατάσταση. Γιατί η δημοκρατία θεμελιώνεται πάνω στην ελευθερία έκφρασης και στον ελεύθερο τύπο. Χωρίς ελεύθερο τύπο δεν είναι νοητή η δημοκρατία. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι η ελευθερία του τύπου όχι μόνο δεν αποτελεί κίνδυνο για την δημόσια ασφάλεια, αλλά αντίθετα θεωρώ κίνδυνο ακόμα και να ακουστεί η ιδέα ότι θα μπορούσε να περιορίσει κάποιος την ελευθερία του τύπου, διότι στην ουσία τότε αυτή που πληγώνεται είναι η δημοκρατία και η δημόσια ελευθερία. Είναι απαραίτητο να διατηρηθεί η ελευθερία της έκφρασης και του τύπου. Όταν έρχεται εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δηλώνει ότι δυστυχώς θεωρεί ότι δεν έχει κανένα περιθώριο κίνησης, εγώ το αμφισβητώ αυτό. Ακόμα όμως και αν συμφωνήσει κανείς με την ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εξακολουθεί να παραμένει η παραβίαση κατά του άρθρου 7 της ε, Συνθήκης Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Και εκεί μπορεί να λάβει μέτρα και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το άρθρο 7 γίνεται σημαντικό όταν υπάρχει υπόνοια παραβίασης του άθρου 2 της ε, συνθήκης που προασπίζεται την ελευθερία και την δημοκρατία. Δηλαδή αξίες οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε κίνδυνο, προφανώς. Δηλαδή, τι σημαίνουν αυτές οι περιστάσεις στη Ρουμανία, θα βγουν τα τάγκς, όχι. Πρόκειται όμως για την υπόνοια παραβίασης του άθρου 7 με αποτέλεσμα ότι θα πρέπει να αρχίσουν οι διαδικασίες που προλέβει το άρθρο 7, δηλαδή αυτό σημαίνει ε, ορισμό ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων οι οποίοι θα εξετάσουν την κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι και το πρώτο και σημαντικότερο βήμα που οφείλουμε να λάβουμε. Και θα ήθελα και πάλι να ακούσω την θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επ' αυτής της προτάσεως. Ε, επεκταθήκαμε επαρκώς για το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς για να κλείνουμε και να λάβουμε μία απόφαση. Νομίζω ότι αφού ακούσαμε την Επίτροπη και τους αναφέροντες, νομίζω ότι η πρόταση της κυρίας Γκρουνή είναι πολύ σκόπιμη, δηλαδή θα μπορούσαμε να οργανώσουμε μία ακρόαση, να μιλήσουμε για την ελευθερία του τύπου και τα προβλήματα που υπάρχουν ως προς την ελευθερία τύπου στην Ευρώπη. Νομίζω ότι μπορούμε να οργανώσουμε αυτή την ακρόαση και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε κατά αυτόν τον τρόπο μέχρι ότου λάβουμε μία απόφαση, δηλαδή μετά από την ακρόαση. Κύριε Μποστινάρ. Απλώς μια διευκρίνηση λέει ο Μποστινάρου. Αν κατάλαβα καλά, θα παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και θα διεξαχθεί επίσης συζήτηση σχετικά με την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Και στο πλαίσιο αυτό θα συζητήσουμε και την ε, ρουμανική περίπτωση. Αυτό είναι σωστό που κατάλαβα. Γκρουνί. Πράγματι θα θέλαμε να γίνει μια ευρεία συζήτηση για την ελευθερία του τύπου, όμως να κλείσει η αναφορά. Και εάν όντως η συζήτηση για την ελευθερία του τύπου καταδείξει ότι εξακολουθούν να υπάρχουν ανησυχίες, μπορούν να καταθέσουν εκ νέου αναφορά. Για την ώρα όμως σήμερα νομίζω ότι δεν έχουμε, δεν έχουμε τα στοιχεία, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε επαρκή θεμελίωση εγώ θα προτιμούσα λοιπόν να κλείσει αναφορά, να ξεκινήσει μια συζήτηση ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη και βλέπουμε. Ο κύριος Μέγερ. Εγώ δεν είμαι υπέρ του κλεισίματος της ε, αναφοράς. Θα μπορούσε να γίνει μια συζήτηση για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες που έχουν ε, εντάξει σε αυτή την αμυντική στρατηγική τη δυνατότητα να κλείσουν ε, ΜΜΕ από κυβερνητικής ε, πλευράς, από πλευράς κυβέρνησης. Αλλά οπωσδήποτε να μην κλείσουμε την αναφορά. Αυτή η συζήτηση ίσως, δείχνει ότι δεν, ίσως να δείξει ότι δεν είναι μόνο μία η περίπτωση παραβίασης όπως η ρουμανική κυρία Άουκεν για ένα λεπτό. Διότι άνοιξε μία συζήτηση με βάση την πρόθεση του και η ρουμανική κυβέρνηση θέλει να απαντήσει. Να δώσουμε το λόγο στη ρουμανική κυβέρνηση. Η κυρία Άουκεν. Η κυρία Άουκεν. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι είναι άσχημη ιδέα να κλείσει η αναφορά. Το θέμα είναι πολύ σοβαρό δεν έχουμε και απάντηση από την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δε κ. Σέφνερ έθεσε ξεκάθαρα ερωτήματα σχετικά με την συνθήκη. Και δεν έχουμε αποφασίσει ακόμη να κάνουμε τη συζήτηση για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το Λαϊκό Κόμμα προσπαθεί να κλείσει αναφορές κάθε, κάθε φορά που του φαίνεται επικίνδυνη μια αναφορά. Χρειαζόμαστε απαντήσεις και πρέπει να συνεχίσουμε γιατί η, η, η αναφορά αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική. Το λόγο δίνω στον κύριο Μπόγκταν Μανίου. Εκπροσωπώ τον Υπουργό Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και εκπροσωπώ και τον πρόεδρο της Ρουμανίας. Θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Στην ε, ε, αμυντική στρατηγική θα ήθελα να πω ότι δεν υπάρχει κανένας ε, τέτοιος περιορισμός και αυτή η κατάσταση ανέκυψε σε σχέση με πολλές ενώσεις δημοσιογράφων. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες δημοσιογράφοι και εδώ την αναφορά την, προώθησαν μόνο μερικές ενώσεις δημοσιογράφων. Ο κύριος Μάιερ έχει δίκιο όταν λέει ότι θα πρέπει να κρίνουμε το... την κάθε αναφορά κατά περίπτωση. Γιατί ε, λέτε ότι στην ε, Ισπανία μόνο η δικαστική αρχή μπορεί να κλείσει μια έκδοση. Εγώ μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν ε, δικαστικές αποφάσεις αλλά δεν έχουν κλείσει ποτέ ε, εκδόσεις, μια έκδοση. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έχασε μια δίκη με τους ε, δημοσιογράφους και αυτό καταδεικνύει την πλήρη ελευθερία που υφίσταται στη Ρουμανία από αυτή την άποψη. Μόνο μία μία ε, κατάσταση της αγοράς, μάλλον μία κακή οικονομική κατάσταση θα μπορούσε να κλείσει μία εφημερίδα ή μία έκδοση, όχι μία δικαστική απόφαση. αυτός που μπορεί να διορθώσει αυτήν την κατάσταση δεν είναι ούτε η κυβέρνηση ούτε το κράτος αλλά μόνο ο ίδιος ο τύπος μπορεί να σταματήσει με αυτή την κατάσταση διαρκούς σπήλωσης. Ευχαριστώ. Perfetto. Per una replica un minuto al petente, poi do la parola alla Commissione, poi formuliamo Λοιπόν, Κομισιόν και μετά θα διατυπώσουμε την πρόταση. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Απλώς μια ε, παρατήρηση ως προς τη διαδικασία. Ακούσαμε τα επιχειρήματα των ΜΕΝ και των ΔΕ και παρά να επιλέξουμε μαζί του να οργανώσουμε μια συζήτηση για την ελευθεροτυπία. Εγώ με τις γνώμες ότι το να μην κάνει κανείς επιλογή είναι και αυτό μια επιλογή και είναι λεπτή η υπόθεση διότι είναι μια αναφορά που έχει υποβληθεί εδώ στην Επιτροπή Αναφορών. Αν πρέπει να έχουμε μια συζήτηση για την ελευθεροτυπία υπάρχει μια Επιτροπή Πολιτισμού, μια Υποεπιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υπάρχει τα μέσα ενημέρωσης, υπάρχει... Ε, δεν είναι καλή αυτή η επιλογή. Uh, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ όλους για τα σχόλια, μερικές διευκρινήσεις δεν είναι ότι δεν παίρνουμε στα σοβαρά το θέμα αυτό, δεν έχουμε αρκετό χρόνο να το αναλύσουμε. Το παίρνουμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα. Όπως το είπε και η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ εδώ, ανησυχούσε για το θέμα, το είπε και την παραθέτω. Η Επιτροπή λέει ότι είναι μια ευκαιρία, ο τύπος δεν είναι μια απειλή και βλέπουμε τη μεγάλη ανησυχία που προκαλεί το θέμα αυτό. Από νομικής απόψεως τα πράγματα είναι σαφή πρέπει να πω. Ε, το θέμα της ανάθεσης αρμοδιοτήτων είναι, περιλαμβάνεται στη συνθήκη και η Επιτροπή δεν μπορεί να κάνει τίποτα από το να επαναλαμβάνει κάθε φορά που δεν έχει αρμοδιότητες, κάθε φορά που είναι εθνικό θέμα, δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε, να παρέμβουμε. Και οι επιπτώσεις της εθνικής στρατηγικής πάνω στην ε, ελευθερία έκφρασης είναι ένα εθνικό θέμα. Βεβαίως, λυπούμεθα ε, η Αντιπρόεδρος Ρέντινγκ εξέφρασε την γνώμη της Επιτροπής, αλλά από νομικής απόψεως η νομοθεσία είναι νομοθεσία και δεν είναι μέσα στις αρμοδιότητές μας να παρεμβαίνουμε για τέτοια θέμα. Η παρέμβαση θυμαίνει ότι αν θέλετε η Κομισιόν να εξετάσει το θέμα αυτό για να αρχίσει μια διαδικασία επί παραβάση, εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι και αυτό ε, προβλέπεται στη συνθήκη της Λισαβόνη για το άρθρο 7 δεν μπορώ να σας δώσω μια οριστική γνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρους όλης της Επιτροπής, αλλά το άρθρο 7 είναι η τελευταία προσφυγή, το τελευταίο ένδικο μέσο το οποίο υπάρχει. Δεν νομίζω ότι υπάρχει το κατόφλι, ότι έχει ξεπεραστεί το κατόφλι σοβαρότητας για να εφαρμοστεί το άρθρο 7. Ευχαριστώ πολύ. το λόγο. Όχι. Εφόσον δεν έχουμε αρμοδιότητα, ζητάω να ψηφίσουμε για το ε, κλείσιμο, αν θέλετε, της αναφοράς. Για τη συζήτηση είναι σαφή τα πράγματα, αποδίδω σημασία και εδώ θα μπορούμε να δούμε μέσα στην Ευρώπη, σε όλα τα κράτη-μέλη, ακόμα και στη Ρουμανία, ακόμα αν υπάρχει μια παραβίαση δικαιωμάτων. Κολέγα Εφνερ. Ναι, σας παρακαλώ όμω να είστε πάρα πολύ σύντομοι, παρακαλώ. Πάρα πολύ σύντομα και σε σχέση με την διαδικασία έθεσα σχετικά με το άρθρο 7 μια ερώτηση και η Επιτροπή απήντησε ότι δεν είχε αρκετό χρόνο για να εξετάσει το θέμα αυτό. Το καταλαβαίνω. Είμαι πλήρη κατανόηση ε, για το θέμα αυτό, αλλά θα ήθελα η Κομισιό να αναλύσει το θέμα, διότι αντίθετα από την Κομισιό είμαι τη γνώμη ότι δεν πρόκειται για παραβίαση εθνικού δικαίου, οπότε τότε δεν μπορούμε να ασχοληθούμε, αλλά παραβίαση του, του ευρωπαϊκού δικαίου. Αν η Κομισιό δηλώνει ότι δεν είχε αρκετό χρόνο ε, για να συμφωνήσει εσωτερικά, τότε η Κομισιόν απλώ χρειάζεται περισσότερο χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε σήμερα να κλείσουμε την αναφορά. Ο κύριος Ποσινάρο. Νομίζω ότι για να υπάρχει αγαστή συνεργασία των μελών αυτής της Επιτροπής και για να μην έχουμε συγκρουσιακές ε, σχέσεις, σας υπενθυμίζω ότι τέσσερις πολιτικές ομάδες ζήτησαν να παραμείνει ανοιχτή αυτή η αναφορά. Δεύτερο, εάν φτάσουμε σε μια κατάσταση ψηφοφορίας, τότε μπορούν να ψηφίσουν μόνο τα μέλη της Επιτροπής και τα αναπληρωματικά μέλη που έχουν κοινοποιήσει τα ονόματά τους μία ώρα πριν στη γραμματή. Όπως είπαμε σήμερα στους συντονιστές, μπορούμε να αναβάλουμε την απόφαση κατά την προσεχή συνεδρίαση, αλλά επαναλαμβάνω την ειλικρινή πρότασή μου. Οι σοσιαλιστές, οι πράσινοι, οι φιλελεύθεροι και οι γκουε ζητάμε να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να γίνει αυτή η συζήτηση για την ελευθερία του τύπου στην Ευρώπη. Το να κλείσει η αναφορά είναι κάτι το απαράδεκτο και είναι σαν να απαξιούμε την εργασία αυτής της Επιτροπής. Ο κυρίως Σαλαφράγκα και μετά θα πρέπει να κλείσουμε τη συζήτηση. Υπάρχουν και άλλες... Θα ήθελα να αναφερθώ στον κανονισμό που όλοι γνωρίζουμε, ξέρει πώς, ε, αναφέρει πώς γίνεται η ψηφοφορία. Εγώ προσπάθησα να σας πω και να το διαβάσει αν θέλει η γραμματεία. Το οποιοδήποτε κάθε μέλος μπορεί να ψηφίσει τη στιγμή που η πολιτική ομάδα ορίσει το ποιες, ποιοι μπορούν να ψηφίσουν και αναπληρώνουν ένα τακτικό μέλος. Θα ήθελα να διαβάσετε τον κανονισμό για να μην υπάρχει καμία... Η συνάδελφος Παλιαδέλη. Απλώς μια πρόταση ε, σχετικά με δύο. Είναι δυνατόν να κρατήσουμε ανοιχτή την αναφορά μέχρι όταν έχουμε την τελική απάντηση της Επιτροπής σχετικά με το άρθρο 7 που ο κύριος Χέφνερ ανέφερε. Θα πρότεινα λοιπόν να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά, όχι με ψηφοφορία μέχρι ότου να περιμένουμε ε, να μας δώσει την απάντησή της η Επιτροπή για το άρθρο 7. Ναι, σας ε, κάνω έκκληση ε, στο αίσθημα υπευθυνότητα που έχετε. Δεν μπορούμε να αφιερώσουμε όλο το πρωινό σε αυτή την αφορά. Σα δίνω τον λόγο, κυρία Νικολάη, αλλά πάρα πολύ σύντομα η Κομισιόν θέλει και αυτή να λάβει τον λόγο πάντοτε σχετικά με την αναφορά αυτή. Εμείς ως φιλελεύθεροι θέλουμε να μείνει η αναφορά ανοιχτή. Νομίζω ότι η ε, η Κομισιόν μας έδωσε μία απάντηση. Δεν μπορούμε να κλείσουμε μία αναφορά κατά αυτόν τον τρόπο. Και τη στιγμή που παραβιάζονται θεμελιώδη δικαιώματα δεν μπορεί να κλείσει αυτή η αναφορά. Θα ήταν πολύ ενοχλητικό. Η Επιτροπή για ένα λεπτό. Ένα λεπτό στην Επιτροπή. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Να υπάρχει μια μικρή παρεξήγηση. Δεν είπα ότι δεν είχαμε αρκετό χρόνο για να αναλύσουμε την αναφορά αυτή. Είπα ότι δεν έχουμε εδώ την εντολή να μιλήσω εκ μέρου της Κομισιόν σχετικά με το άρθρο 7. Η γνώμη μου είναι ε, και αυτό νομίζουμε στην Κομισιόν ότι το θέμα αυτό ε, δεν υπερβαίνει το κατόφλι ε, το οποίο απαιτείται το κατώτατο όριο για την εφαρμογή του άρθρου 7. Δεν είναι μέσα στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων μας, δεν είναι θέμα χρόνου, οι θέσεις είναι σαφές ότι δεν πρόκειται για ένα θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λοιπόν, η κατάσταση ε, δεν είναι απλή όπως βλέπουμε, αλλά μου φαίνεται σαφές ότι η Επιτροπή δηλώνει ότι δεν είναι αρμόδια, είναι αναρμόδια. Αυτό λέχθηκε ρητά. Και τώρα μια υπενθύμηση διαδικαστική. Υπάρχει ένα αίτημα για ψηφοφορία. Υπενθύμηση κανονισμού. Και μπορώ να πω ότι το παράγραφος 2 του άρθρου 147 σχετικά με τους αναπληρωτές λέει ότι το μέλος σε περίπτωση απουσίας ενός μέλους της Επιτροπής αν δεν υπάρχει διορισμός ενός μονίμου αναπληρωτή αντικαταστάτη θα πρέπει το όνομα του αντικαταστάτη να αναφέρεται πριν την έναρξη της ψηφοφορίας. Είναι σαφές λοιπόν ότι η παρουσία ε, ισοδυναμεί με ανακοίνωση είναι κάτι το που υπονοείται. Κάτι το αυτονόητο. Βεβαίως αυτή η Επίτροπη δεν έχει τη συνήθεια να ψηφίζει. Είναι μια Επιτροπή στην οποία δεν επιτυγχάνουμε ίσως, αλλά όπου θα έπρεπε να εφαρμόζουμε ε, την πολιτική με αμερόληπτο τρόπο, χωρίς μεροληψίες και υπερβολές. Διότι αυτή είναι η χρησιμότητά μας και σε αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση όπου είναι προφανές ότι υπάρχει κάτι το επίμαχο τώρα, ένα επίμαχο θέμα το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μια ψηφοφορία όπου θα λάβουν μέρος οι παρόντες διότι είμαστε υποχρεωμένοι να λάβουμε αυτού του είδους ε, την απόφαση, αυτό διότι αυτό προβλέπεται από τον κανονισμό. Αν ε, υπάρχει ένα αίτημα για ψηφοφορία, ε, είναι, πρέπει να ψηφίσουμε για τις προτάσεις. Συνήθως αυτό γίνεται με άτυπο τρόπο, αλλά εδώ... Λοιπόν, Τώρα πρέπει να σας δώσω τις ανακοινώσεις σχετικά με τους αναπληρωτές και αντικαταστάτες. Θα ήθελα να ε, περιμένετε λίγο κύριε Μποσινάρο, δύο λεπτά, όχι παραπάνω. Σας δίνω αυτά τα δύο λεπτά, αλλά δεν ξέρω. Θέλετε να αναφέρω ονομαστικά όλους τους αναπληρωτές. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι απαραίτητο. Το έγγραφο το οποίο υποβλήθηκε στην Προεδρία υπάρχει και υπάρχει μια πρόταση για να κλείσουμε την αναφορά και να, τη, να παραπέμψουμε ενδεχομένως τους συντονιστές. Αγαπητοί συνάδελφοι, ας χρησιμοποιήσουμε ωφέλιμα ε, τα δύο λεπτά. Να κλείσουμε λοιπόν, η πρόταση είναι να κλείσουμε την αναφορά ε, και να υποβάλλουμε στην διάσκεψη των συντονιστών ε, το αίτημα για να οργανωθεί ένα, μια συζήτηση για να ελευθεροτυπία στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν και την πρόταση της άλλης ομάδας λοιπόν ε, να αφήσουμε ανοιχτή την αναφορά περιμένοντας την απάντηση της Κομισιό. Αλλά μας δόθηκε τώρα η απάντηση της Κομισιό. S'il Sí. Colega, eh, Presidenta, eh, por favor. On Presidenta, por favor. Sí, sí, perdón. Si vamos, si vamos... Momento. Un momento. Allora, riprendiamo. Ένα λεπτό. Λοιπόν, τώρα συνεχίζουμε τις εργασίες μας. Σας παρακαλώ. Εάν είναι να, ψηφίσουμε, ας ψηφίσουμε αμέσως, γιατί υπάρχουν και άλλες αναφορές. Ας γίνει αμέσως, διότι ήδη έχουμε μία ώρα καθυστέρηση. Ναι, μου ζητήθηκαν δύο λεπτά. Ο κύριος Κάσμου. Ε, Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δεν ε, είμαι εντεταλμένος να μιλήσω, αλλά έχω κάποια πείρα ως αντιπρόεδρος αυτής της Επιτροπής επί πέντε χρόνια. Δεν υπάρχει προηγούμενο να ψηφίσουμε χωρίς την συμφωνία όλων των πολιτικών κομμάτων και χωρίς προηγούμενη ανακοίνωση ε, στα κόμματα. Για να υπάρχει ψηφοφορία θα πρέπει να περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη και είναι μέρος της ε, διαδικασίας και των ε, προηγουμένων ότι όταν υπάρχει ένα μέλος που αποφασίζει να μείνει ανοιχτή μια αναφορά θα πρέπει η αναφορά να μείνει ανοιχτή εάν προβούμε σε ψηφοφορία ή όχι. Θα σας πω ότι η ομάδα μου δεν θα ψηφίσει, διότι πιστεύουμε ότι δεν υπάρχει προηγούμενο για μια τέτοια ψηφοφορία. Είναι αντισυνταγματική αυτή η ψηφοφορία. Θα την αμφισβητήσουμε εφόσον υπάρχουν τα προηγούμενα. Έχω την εμπειρία 7 ε, ετών σε αυτή την Επιτροπή και θεωρούμε ότι ε, δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο δεν είναι μόνο η ομάδα μου, αλλά νομίζω και άλλες ομάδες θα σκεφτούν ότι δεν είναι ακατάλληλη αυτή η ψηφοφορία και λοιπόν σας ζητώ να μην προβούμε σε ψηφοφορία. Υπάρχει ακόμα μια αίτηση λήψεως του λόγου. Η Τουργκάης παρακαλώ. Όπως είπε ο ίδιος ο κ. Κάσμαν, Έχει δίκιο βέβαια. Όταν μια πολιτική ομάδα επιθυμεί να διατηρηθεί ανοιχτή η αναφορά, αλλά για την Κύπρο για παράδειγμα είχε η δική του ομάδα πάλι ζητήσει να παραμείνει ανοιχτή αναφορά τελικά όμως κάναμε ψηφοφορία αλλά στην επόμενη, στην επόμενη ε, συνεδρίαση όμως πρέπει να εγγραφεί στην ημερήσια διάταξη η, η ψηφοφορία. Ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τα όργανα λαμβάνουν αποφάσεις με πλειοψηφία. Είμαι συντονιστή στην Επιτροπή Εξωτερικών και όπως ξέρει και ο κύριος Μάιερ που είναι συντονιστής λαμβάνονται από ε, το θεσμικό όργανο. Όταν μια πολιτική ομάδα ζητεί να γίνει μια ψηφοφορία, οφείλει να εκτελείται αυτή η ψηφοφορία. Δεν μπορεί να ανακόπτεται η διαδικασία όταν βλέπει κάποια ομάδα ότι θα χάσει την ψηφοφορία. Έτσι λειτουργούν τα δημοκρατικά όργανα. Κυρία Πρόεδρε, παρακαλώ να εφαρμόσετε τον κανονισμό και παρακαλώ τις συναδέλφους και τους συναδέλφους με να δείξουν τον ίδιο σεβασμό που έδειξα και εγώ και άκουσα όλες τις παρεμβάσεις, να ακούσουν λοιπόν και την δική μου. Όταν μια πολιτική ομάδα επικαλούμενη την, τον κανονισμό ζητεί να γίνει ψηφοφορία, οφείλει να εκτελείται η ψηφοφορία. Δεν ψηφίζουν οι συντονιστές, ψηφίζουν τα μέλη της Επιτροπής που έχουν δικαίωμα ψήφου. Και μου φαίνεται αντιδημοκρατικό όταν μια πολιτική ομάδα βλέπει ότι δεν έχει στη διάθεσή της επαρκή μέλη να ζητεί να αναβάλλεται η, ψηφοφορία. η ψηφοφορία. Συγγνώμη. Παρακαλώ να προχωρήσετε σύμφωνα με αίτηση του Λαϊκού Κόμματος σε ψηφοφορία. Μέγερ, τελευταίος. Κυρία Πρόεδρε, εγώ θα απευθύνω έκκληση στους συναδέλφους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος ότι ο ίδιος ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είπε ότι δεν έχει εντολή σύμφωνα με το άρθρο 7 για το άρθρο 7 μάλλον δεν έχει και επειδή και άλλες πολιτικές ομάδες είπαν ότι υπάρχει ενδεχόμενο παραβιάσεως του άρθρου 7. Ας αναβάλουμε το θέμα και ας το επανεγγράψουμε στην ημερήσια διάταξη. Νομίζω ότι είναι λογικό να το πράξουμε. Ακούσαμε τις απόψεις των κοινοβουλευτικών ομάδων εδώ, ακούσαμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που λέει ότι δεν έχει εντολή για να εξετάζει θέματα παραβιάσεως του 7. Ας γίνει ψηφοφορία λοιπόν την επόμενη συνεδρίαση. Θα δώσω το λόγο σε όλους, αλλά έχουμε και άλλες, ε, και άλλες αναφορές. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε ε, πάπυρον. Ζανούκα, Πρέντα και μετά Αρκή. Σας ευχαριστώ. Φαίνεται πως το Λαϊκό Κόμμα δεν θέλει να γίνει ψηφοφορία όταν είναι μόνοι τους. Ε, αλλά δεν θα έχετε όμως απαρτία εάν ψηφίσετε μόνοι σας χωρίς τους υπολείπους, χωρίς τις υπόλοιπες κοινοβουλευτικές ομάδες. Εύκολη λύση αλλά όχι δημοκρατική. Αν θέλετε να λήξετε την υπόθεση αυτή δεν συμμετέχουμε εμείς και μόνος δεν έχετε απαρτία. Ο κύριος Πρέντα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά με ευνηδιάζουν λίγο οι εξελίξεις. Αρνούνται ορισμένες ομάδες την, ε, την ενέργεια ψηφοφορίας. Δεν έχω μεγάλη ε, εμπειρία στην Ευρωβουλή, αλλά πώς είναι δυνατόν να περιφρονούν την βούληση μιας πολιτικής ομάδας. Ωραία, ορισμένοι είναι απόντες. Εντάξει, ίσως ε, δεν μπόρεσαν να προσέλθουν λόγω χιονοπτώσεων. Αλλά ας γίνει ψηφοφορία, είναι απλό. Αν όμως προσπαθούν να παρακολουθήσουν την ψηφοφορία, αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού και απέναντι στους ίδιους αναφερόμενους, οι οποίοι περιμένουν απάντηση από μας. Η Πρόεδρος. Επ' αυτού, νομίζω ότι χρειάζεται να ισχύσει μια κοινή λογική πράγματι, αλλά υπάρχουν και οι κανονισμοί που οφείλουμε να σεβαστούμε. Αν μπορούμε να συμφωνήσουμε μεταξύ των πολιτικών ομάδων ότι θα κάνουμε το σύνηθε, διότι αλλιώ αν δεν υπάρξει τέτοια συμφωνία δεν μπορώ να κάνω τίποτε άλλο παρά να ε, εκτελέσω ψηφοφορία, να διενεργήσω ψηφοφορία. Κύριε Κάσμαν, ε, απευθύνομαι και στην δική σας πείρα. Ε, διδάσκομαι από τη δική σας πείρα ασφαλώς, αλλά επιτρέψτε μου να πω ότι έστω και ανεπίσημα θα ψηφίσει η Επιτροπή. Διότι στο τέλος της συζητήσεως ε, θα ρωτήσω τους συναδέλφους να δηλώσουν τι επιθυμούν να πράξουν. Η απόφαση λαμβάνεται από την ολομέλεια της Επιτροπής. Εάν δηλαδή θα κλείσει η αναφορά, θα παραμείνει ανοιχτή Το ίδιο ψηφοφορίες γίνονται και για άλλα θέματα. Το μόνο που μπορώ να κάνω λοιπόν είναι να διενεργήσω ψηφοφορία. Η αίτηση ψηφοφορίας λοιπόν από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα επιβεβαιώνεται και αυτό γίνεται και συνήθως. Αν θέλετε θα ζητήσουμε από την νομική υπηρεσία να μας πει ε, εάν είναι ορθό αυτό. Έχουν ζητήσει λοιπόν κατεπανάλη ψηφοφορία και υποχρεωμένοι να την διεξαγαγώ. Ε, ο κ. Κάσμαν, επιτρέψτε μου Κύρια Πρόεδρε, επειδή απευθυνθήκατε σε μένα, είπατε ότι η Ολομέλεια της Επιτροπής μπορεί να αποφασίσει. Εάν κλείστε την ε, αναφορά, ωστόσο, δεν μπορεί να αποφασίσει η Ολομέλεια της Επιτροπής, γιατί δεν θα προχωρήσει η αναφορά. Δοθέντως ότι το Λαϊκό Κόμμα είναι η μόνη πολιτική ομάδα που θέλει να ψηφίσει. Εγώ θα υποστηριξώ ότι εφόσον προχωρήσει την ψηφοφορία, οι πολιτικές εκείνες ομάδες που δεν επιθυμούν να συμμετάσχουν στην ψηφοφορία θα αποχωρήσουμε και θα επανέλθουμε όταν θα έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία. Διότι θεωρούμε ότι η απόφαση αυτή, εφόσον ληφθεί, θα αμφισβητηθεί ενώπιον της διασκέψη των Πρόεδρων. Αυτό ήδη προανακοινώθηκε. Εν πάση περιπτώσει, εφόσον διατυπώθηκε το αίτημα, δεν μπορώ να το απαρνηθώ. Κύριε Σαλαφράγκα, μόνο αν πρόκειται για ένα συμφιλιωτικό θέμα, διότι ξέρουμε τον κανονισμό. Επειδή είπατε ότι μπορεί να παραπεμφθεί το θέμα στη διάσκεψη των ε, Προέδρων, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το άρθρο 195 παράγραφος 2. Λέει ότι ισχύει η ψηφοφορία στην Επιτροπή εάν είναι παρόν το 1 τέταρτον των μελών. Άρα το θέμα είναι απόλυτα σαφές. Η συντονίστρια της ομάδας μου ζήτησε να διεξαχθεί η ψηφοφορία και χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση ζητώ να διεξαχθεί. η κυρία Γκρουνή προτείνει να κλείσουμε την αναφορά και να γίνει μια συζήτηση για την ελευθερία τύπου στην Ευρώπη και ενδεχομένως να διοργανωθεί μια κρόε. E Αρχίζει η ψηφοφορία. Apro la votazione sulla proposta formulata dalla eh, Λοιπόν, πρόταση συγκρουνή. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης Γκρουνή. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η πρόταση. Ωραία, ας γίνει η καταμέτρηση. Παρακαλώ η γραμματεία να κάνει την καταμέτρηση.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 ψήφισαν 15 υπέρ με την αποχή της Προέδρου, άρα κλείνει η αναφορά.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 Ωραία σας. Ας επανέλθουμε στις εργασίες μας εντάχει. Ζητώ συγγνώμη από τους αναφέροντες. Σημείο 18 και σας ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Δίνω το λόγο στον αναφέροντα. 587 του 2008. Ο κύριος Φερνάντες ε, έχει το λόγο. Φουάρος, Φερνάντες Φουάρος. Δεν ξέρω κατά πόσο θα πρέπει να αρχίσω πριν προσέλθουν και οι υπόλοιποι γιατί έφυγαν από την αίθουσα. Να περιμένουμε λίγο. Όχι, να αρχίσετε. Ε, ε, Θα ήθελα να περιμένω να επανέλθουν και τα υπόλοιπα μέλη βουλευτέ στην αίθουσα. Υπάρχει επαρκή αριθμό. Ε, για να επανέλθουμε. Σας παρακαλώ να επανέλθετε, διότι ήδη έχουμε υπερβεί κατά πολύ το χρόνο μας. Muy Señora Presidenta. Πρόεδρε, μέλη της Επιτροπής σας ευχαριστώ γιατί μας δίνετε τη δυνατότητα να παραθέσουμε τα επιχειρήματά μας. Θέλουμε να κυρωθεί η καταγγελία του Μαρτίου του 2009. Σύμφωνα με την έκθεση Επιτροπής Περιβάλλοντος, η κυβέρνηση Ισπανία και των Καναρίων νήσων θεώρησαν ότι το παρατηρητήριο περιβάλλοντος Puerto de Granadilla δημιουργήθηκε για την προστασία του περιβάλλοντος και να επιβληθούν τα σωστά και αντισταθμιστικά μέτρα. Δυστυχώς όμως δεν πληρώθηκαν αυτοί οι στόχοι και η Επιτροπή θα πρέπει να λάβει επαρκώς υπόψη την κατάσταση αυτή. Καταρχήν ο διορισμός του Διευθυντού του Ιδρύματος παραβαίνει την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία διότι διορίστηκε άμεσα χωρίς τις εγγυήσεις που ορίζει ο νόμος. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με το ψήφισμα του περί Ευρωπαϊκών Ιδρυμάτων 304 κάθετος 93 και τον ε, νόμο 50 κάθετο, 2002 της 26 Δεκεμβρίου για τα ε, δημόσια ιδρύματα ορίζει στο άρθρο 46 ότι η επιλογή του προσωπικού θα πρέπει να λάβει χώρα με βάση συνθήκες ισονομίας, αξιοκρατίας, και προσόντων, σύμφωνα με τη, τους όρους του διαγωνισμού. Επίσης, η συμβατική σχέση θα βασίζεται σε αντικειμενικά κριτήρια, κριτήρια υγιούς άμυλας, έτσι ώστε να μπορούν να προταθούν σωστές προτάσεις, αλλά βλέπουμε ότι αυτό, ε, ο διορισμός αυτός αντιβαίνει σε αυτές τις αρχές. Αυτές οι αρχές δεν τηρήθηκαν διότι διορίστηκε ο διευθυντής της, ε, του Ιδρύματος Puerto de Granadilla άμεσα με συνοπτικές διαδικασίες από την εργοδοσία. Από την άλλη πλευρά, ως προς τα διορθωτικά ε, μέτρα που ορίζει η Επιτροπή, όπως το bypass που θα έπρεπε να πραγματοποιηθεί, δεν έγινε. Σήμερα ούτε καν υφίσταται, δεν έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα και αυτό αφορά και την, το έργο του αναχώματος προστασίας που δεν έχει πραγματοποιηθεί. Ε, μία άλλη τήρηση αφορά ότι η κυβέρνηση των Καναρίων νήσων ε, ε, έβγαλε από τον κατάλογο εκατοντάδες είδη υποπροστασία από τον ε, Εθνικό Κατάλογο που ε, ενυπάρχει και στη συνθήκη του Άρχους που έχει υπογράψει η Ισπανική κυβέρνηση. Αυτή τη στιγμή εκρεμεί η υπόθεση στο Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων. Το ίδιο το δικαστήριο έθιξε ένα θέμα αντισυνταγματικότητας για την παραβίαση του συστήματος κατανομής αρμοδιοτήτων στο κράτος μέλος. Η Επιτροπή θα πρέπει να γνωρίζει ότι άρχισαν τα έργα του Puerto de Granadilla με την εκρεμή αυτή υπόθεση ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου των Καναρίων Νήσων. Χωρίς την έγκριση των εν λόγω έργων από το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Επιτροπή Υποδομών του Λιμένος παραβιάζοντας το άρθρο 38 του νόμου 48 κάθετος 2003 του οικονομικού, ε, του, της οικονομικής πλαισίωσης, του νόμου πλαισίου οικονομικών υποθέσεων και παροχής υπηρεσιών για τους ε, λιμένες γενικού ενδιαφέροντος. Άρα, οι λιμενικές αρχές της Σαντακρούς, της Τενερίφης δεν είναι αρμόδιος οργανισμός για να εγκρίνει την απαρχή των έργων στο Πουέρτο Γκραναντίλια. Και όμως ανέθεσε στις ε, ε, ανάδοχες εταιρείες το έργο του αναχώματος, τις δημιουργίες του αναχώματος χωρίς την έγκριση του Υπουργείου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι ένας αυτόνομος οργανισμός. Δηλαδή ότι το Ίδρυμα Παρατηρητήριο που de Granadilla ε, εισακούει τις ε, πολιτικές προσταγές της νήσου. Λαμβάνοντας υπόψη την ε, στάση των λιμενικών αρχών της Σαντα και τις ε, καταγγελίες των οικολογικών οργανώσεων, οι εισαγγελικές αρχές θα πρέπει να αναλάβουν την υπόθεση έτσι ώστε να επιληθεί αυτό το ποινικό αδίκημα οικολογικού χαρακτήρα. Το πρόγραμμα του Puerto de Granadilla έχει ένα προηγούμενο, το Puerto de Arinaga, στις Λασπάλμας ε, της ε, Μεγάλης Καναρίου νήσου και όπως και στην περίπτωση της Γκρανατίγια και εκεί αναλήφθησαν έργα χωρίς να μπορεί να γίνει πολύ σωστά το άδειασμα και η φόρτωση των εμπορευματοκιβωτίων. Και είναι ένα ζήτημα το οποίο εκκρεμεί επίσης το Ανώτατο Δικαστήριο των Καναρίων Νήσων. Επίσης έγινε κα, ε, κατασπατάληση των διαρθρωτικών ταμείων ε, με βάση την προστασία του περιβάλλοντος όπως θα έπρεπε να είχε προωθηθεί κατά το κατασκευαστικό αυτό έργο του Puerto de Granadilla. Έχουν ε, υποβληθεί 16 ερωτήσεις στη Γερουσία σε σχέση με την απομάκρυνση από τον κατάλογο των υποπροστασία ειδών και υπάρχουν ζητήματα ε, παρελκόμενα ζητήματα, δεν έχουν, παρεπόμενα με συγχωρείτε, ζητήματα τα οποία δεν έχουν απαντηθεί μέχρι τούδε. Θα θέλαμε η Επιτροπή σας να ε, δεχτεί να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου επιληθεί το ζήτημα από τα Ισπανικά δικαστήρια να ζητηθεί από την Επιτροπή να εποπτεύσει και να επαληθεύσει τα δεδομένα με ανεξάρτητη έρευνα. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν δέχομαι άλλες συζητήσεις. Δυστυχώς παρακολύεται το, το έργο μας και την παρουσίαση του αναφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Απλώς θα ήθελα να πω ότι για ζητούμε με βάση τα ανωτέρα η Επιτροπή να επιτρέψει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά μέχρι ότου επιληθεί το ζήτημα από τα δικαστήρια της Ισπανίας, τα Ισπανικά δικαστήρια και δεύτερον να ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επαληθεύσει τα οσάνο εκτεθέντα με μία ανεξάρτητη έρευνα σε σχέση με την απομάκρυνση από τον κατάλογο των υποπροστασία ειδών και αυτό να γίνει από μια ανεξάρτητη επιτροπή. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Ανοίγει η συζήτηση. Δίνουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Επιτροπής. Muchas gracias, señor presidente. En a la presencia de los peticionarios, me Θα ήθελα να μιλήσω κι εγώ στα ισπανικά. Υπάρχουν διάφορες πτυχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον σε αυτή την αναφορά. Όπως ξέρετε, οι κατασκευαστικές, ε, τα κατασκευαστικά έργα στο που de ε, σχετίζονται και με άλλα κατασκευαστικά έργα που είχαν προϋπάρξει και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο υπάρχει συμμόρφωση ως προς την ε, τρέχουσα νομοθεσία της, ε, στην ε, χώρα αυτή, στην Ισπανία. Και θεωρούμε ότι επειδή αφορά την εσωτερική ένομη τάξη, εμείς δεν μπορούμε να παρέμβουμε. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο τηρείται σωστά η κοινοτική νομοθεσία σε σχέση με αυτή την νομοθεσία θυμόσαστε ότι όσον αφορά το Puerto de Granadilla, ε, υπαγόταν στο άρθρο 6 ε, με βάση την οδηγία 43 του 83 σε σχέση με την προστασία της χλωρίδας και της πανίδας και έγινε μία ανταλλαγή πληροφοριών με τις, υπηρεσίες, με τις υπηρεσίες της ε, Επιτροπής, όχι μόνο με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος, αλλά και με άλλες γενικές διευθύνσεις που ήταν αρμόδιες. Στις 2006 συντάχθηκε η γνωμοδότηση της Επιτροπής και δυνάμει του άρθρου 6.4 που ανέφερα, που προανέφερα, αναφέρονται οι όροι και οι συνθήκες που πρέπει να διέπουν την κοινοτική περιβαλλοντική νομοθεσία. Το δεύτερο σημείο είναι ποια ήταν η θέση της Επιτροπής όταν ελήφθη από αυτή η απόφαση. Δηλαδή μας ενδιαφέρει η συμμόρφωση στη γνωμοδότηση της Επιτροπής Δεν μπορούμε όμως να αγνοήσουμε το εξής, ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των Καναρίων Νήσων που είναι η αναστολή. Γι' αυτό θα πρέπει το Ανώτατο Δικαστήριο να απόφανθει και τη στιγμή που ανεστάλλει η απόφαση δεν θα ήταν σκόπιμο να αποφανθεί η Επιτροπή προγενέστερα. Υπάρχει και μία άλλη πτύχη. Δηλαδή, μέσα στα πλαίσια αυτής της αναστολής δεν θα πρέπει να εκτελούνται τα έργα. Και βλέπουμε ότι κατά αυτόν τον τρόπο τηρείται η γνωμοδότηση. Ως προς τα επαπειλούμενα είδη υπάρχει η νομοθεσία των Καναρίων νήσων. Το περιεχόμενο δεν είναι απόλυτα σαφές, γι' αυτό η Επιτροπή αυτή τη στιγμή ερευνά το ζήτημα για να διευκρινιστούν οι αμφίβολες πτυχές αυτές της νομοθεσίας που αφορά τα προστατευόμενα είδη. δεν μπορούμε να ε, δράσουμε σε αυτό το, το, τη δεύτερη πτυχή, το δεύτερο σκέλος του ερωτήματος σε σχέση με τα επαπειλούμενα είδη. Θα θέλαμε περισσότερες ε, πληροφορίες. Και θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε γιατί επισκεφτήκατε τη Γενική Διεύθυνση Ρέτζιο και την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος για να διευκρινίσετε αυτό το δεύτερο ε, σκέλος ε, παρέμβασης, δηλαδή σε σχέση με τα επαπειλούμενα είδη. Και με συνοδεύει και η αρμόδια που μπορεί να σας μιλήσει για αυτό το δεύτερο σκέλος. Σας ευχαριστώ πολύ για την πληροφόρηση. δίνω το λόγο στην αρμόδια της Επιτροπής. Θα προσθέσω μόνο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή η κατάσταση, πώς προχωρεί αυτό το έργο του Πουέρτο Γραναδία. Ε, δεν προχωρεί, έχει διακοπεί δεν <clears throat> δόθηκε χρηματοδότηση από πλευρά Ευρωπαϊκή Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τον Μάρτιο του 2009 η χώρα μέλος δια των διοικητικών αρχών της υπέβαλε πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αίτηση χρηματοδότησης. Τον Απρίλιο του 2009 η υπηρεσία της Κομισιόν θεώρησαν παραδεκτή την αίτηση αυτή, σύμφωνα με τους δικείους κανονισμούς. Τον Μάιο του 2009 έγινε η διακοπή της ε, περαιτέρω κατασκευής του έργου. Μέχρι ότου αποσαφινιστούν οι νομικές πτυχές του θέματος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Εκεί βρίσκεται η κατάσταση σε ό,τι αφορά αυτό το έργο. Σας ευχαριστώ. Εδώ και πέντε χρόνια, όταν ήμουν πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου των ε, Καναρίων Νήσων, είχα προβάλει μία παρόμοια αναφορά που εκπροσωπεί 2 εκατομμύρια κατοίκους και υπήρχε ε, ομοφωνία όλων των κατοίκων. Δηλαδή εκπροσωπούμε 2 εκατομμύρια κατοίκους των Καναρίων νήσων. Και πιστεύω και δέχομαι τις διάφορες απόψεις που προβάλλονται. Επαναλαμβάνω την ελπίδα μου να προβάλλουμε ε, αυτή την υποδομή που είναι πολύ σημαντική και για τα Κανάρια νησιά και για όλο, ολόκληρη την Ευρώπη. Πέντε χρόνια μετά βλέπουμε ότι μερικοί καταβάλουν προσπάθειες έτσι ώστε αυτό το έργο να παρακολουθεί. Δεν υπάρχει καμία, κανένα αποδοκτικό στοιχείο, δεν υπάρχει καμία νομική ή επιστημονική βάση η οποία να μην έχει ληφθεί είτε στον επιστημονικό τομέα όσο και στον νομικό. Εγώ σέβομαι τον αναφέροντα, αλλά αναμειγνύει πολλά πράγματα. Νομίζω ότι θα πρέπει να αρκεστούμε στην αναφορά και όχι στην εκτέλεση του, του προγράμματος. Δηλαδή αναμειγνύει την υποδομή, μιλάει για το παρατηρητήριο, μιλάει για το διορισμό του διευθυντή, μιλάει για την υποστήριξη από τα Κανάρια, από την κυβέρνηση των Καναρίων νησιών, δηλαδή αναμειγνύει το έργο το ίδιο, την υποδομή, το διορισμό του διευθυντή ενώ αυτό που μας ενδιαφέρει είναι κατά πόσο το παρατηρητήριο αυτό είναι ανεξάρτητο ή όχι. Αναμειγνύει και την Ένωση των Περιβαλλοντικών Οργανώσεων όπου δεν συμμετέχουν οι οικολογικές οργανώσεις που ε, συμμετείχαν κατά των έργων του που έρθονται Γκραναντίγια. Δηλαδή, δεν έχουμε να κάνουμε παρά με μία πρόσμιξη πολλών στοιχείων. Νομίζω ότι ελέγχθη ότι έγινε ένας ε, διορισμός που δεν ακολούθησε δημοκρατική διαδικασία. Δηλαδή, εντάξει, διορίστηκε από την εργοδοσία. Ενώ αναφέρεται στην αναφορά ότι ε, διορίστηκε από τις αρχές. Η αλήθεια όμως είναι ότι διορίστηκε από την εργοδοσία. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι λιμενικές αρχές πρότειναν ε, οι λιμενικές αρχές πρότειναν ορισμένους ε, συγκεκριμένους διορισμούς και τις υποστήριξαν τα πανεπιστήμια καθώς και η Ένωση των Θαλασσίων Πόρων των Καναρίων Νήσων. Ε, εάν δείτε την ιστοσελίδα μας θα δείτε ότι αυτοί οι διορισμοί έχουν δημοσιοποιηθεί πολύ σωστά. Άρα θα πρέπει να αναλύσετε κατά πόσο αυτή η αναφορά αντικατοπτρίζει την αλήθεια, δηλαδή κατά πόσο υπάρχει ανεξάρτητος ε, διορισμός. Στις 31 Μαρτίου του 2009 η Επιτροπή μίλησε για την ανεξαρτησία του παρατηρητήου και είπε ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικοί λόγοι για να αμφισβητήσουμε την νομιμότητα της διαδικασίας διορισμού. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μπορούμε να μιλήσουμε για το ανώτατο δικαστήριο για την παράλυση των έργων. Εδώ και τρεις μήνες το Κοινοβούλιο των Καναρίων Νήσων άλλαξε τον νόμο και άρα ε, τα έργα θα συνεχιστούν, δηλαδή ξεκινάει εκ νέου η διαδικασία. Δεν μπορούμε να αφήσουμε ανοιχτό συνεντίε αυτό το θέμα. Το μόνο θέμα είναι, ε, που θίγεται είναι η ανεξαρτησία του παρατηρητηρίου. Πιστεύω ότι αυτή η Επιτροπή θα πρέπει να προωθήσει αυτό το έργο που είναι ύψης της σημασίας για τα Κανάρια νησιά, για την Τενερίφη και για όλα τα νησιά. Η κυρία Άουκεν. Σύντομα, κύριε Πρόεδρε. Δεν είναι ορθό να λέγεται ότι δεν υπάρχουν προβλήματα όσο δεν έχει αποφασίσει το δικαστήριο. Υπάρχουν προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά και να επιμείνουμε, εάν συνεχιστεί το έργο, τουλάχιστον οι όροι που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει να πληρούνται. Σύμφωνα με αυτά που ακούσαμε σήμερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά περιλαμβάνεται και στα έγγραφά μας, υπάρχουν προβλήματα. Το ανώτατο δικαστήριο των Κανάριων νησιών το έχει επίσης δεχθεί και η Κομισιόν λέει ότι υπάρχουν προβλήματα με τις σχετικές οδηγίες. Κατά συμπέρασμα πρέπει να παραμείνει ανοιχτή η αναφορά. Σας ευχαριστώ κύριε Άουκεν. Η Τουργκάης. Μη μας ε, προκαλείτε πάλι κύριε Άουκεν. Νομίζω ότι είναι η τρίτη φορά που συζητούμε το ίδιο θέμα. Σας υπενθυμίζω όταν ο κύριο Μάρτο ήταν παρόν εδώ ως εκπρόσωπος ε, του Κοινοβουλίου των Καναρίων και μαζί και με άλλες πολλές αρχές των Καναρίων νησιών, τοπικές αρχές κλπ. Και είχαν ζητήσει, είχαν ε, μάλλον δηλώσει την υποστήριξή τους για το έργο αυτό και για όλη την Ισπανία μάλιστα. Είναι λοιπόν ιδιαίτερο το θέμα κυρία Πρόεδρε. Η αναφορά ε, έχει ορισμένα χρόνια στην πλάτη της ήδη. Η κυρία Γιάλα ήταν επίσης παρούσα τότε. Έχουν περάσει χρόνια, αλλά θυμούμαστε όλοι ότι η αναφορά αυτή είχε κλείσει, μετά ξανά άνοιξε, διότι ο εκπρόσωπος των Πράσινων, όπως είπε και η κυρία Άουκεν, είχε νέες πληροφορίες για το ίδιο θέμα και με τα επιχειρήματα εκείνα λοιπόν είχαμε ανοίξει και πάλι την αναφορά για δεύτερη και για τρίτη φορά, όπως έχει λοιπόν σήμερα. Ο κύριος Μάρτο είπε αν δεν υπάρχουν άλλα επιχειρήματα ή θέματα την έχουμε συζητήσει την αναφορά αυτή για τρίτη φορά. Κάποια στιγμή πρέπει να λάβουμε μια απόφαση. Μπορούμε να ψηφίσουμε και εδώ τώρα. Γιατί όπως είπα άνοιξε, έγκλεισε, ξανάνοιξε, ξαναέγκλεισε, τώρα είναι τρίτη φορά. Ακούσαμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δεν υπάρχουν και νέες πληροφορίες. Νομίζω πρέπει να κλείσει πια αν δεν έχουν άλλες. Α, ναι, η κυρία Γκρινή. Απλώς για να επιβεβαιώσω την ε, θέση του συναδέλφου Καρλος Χιταγκός και να ζητήσω να κλείσει αυτή η αναφορά, εφόσον δεν ε, περιμένουμε πλέον συμπληρωματικές πληροφορίες. Εάν δεν υπάρχουν δεν... άλλες παρεμβάσεις, θα ήθελα να πω προς τον κύριο Μάτο ότι ζητήθηκε να κλείσει να κλείσει αυτό το θέμα. Ίσως θα πρέπει να ακολουθήσουμε το πνεύμα που μας διείπε και στην περίπτωση του θέματος της Ρουμανίας. Δηλαδή η Επιτροπή είπε ότι δεν είναι θέμα δικό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπάρχουν όμως άλλα ζητήματα ε, στα οποία ε, για τα οποία ζήτησε επιπρόσθετες πληροφορίες η Επιτροπή σε σχέση με τα υποπροστασία είδη, με τα επαπειλούμενα είδη. Και η Επιτροπή είπε σε σχέση με τις επιδοτήσεις ότι όλα τα έργα έχουν παραλύσει διότι ε, υπάρχει εκκρεμωδικία. Και δεν κατά πόσο με βάση τη, τη λογική που μας δείπε στην περίπτωση της Ρουμανίας δεν θα πρέπει να ψηφίσουμε. Εάν θέλετε να εφαρμόσουμε την ψηφοφορία, κανένα πρόβλημα. Σας είπα όμως τι είπαμε οι τέσσερις ομάδες, ομάδες πριν. Ή θα εφαρμόσετε την ψηφοφορία και αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς οι τέσσερις ομάδες δεν θα αντιταχθούμε. Άρα θα μπούμε σε μία δυναμική που είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Κάνω έκκληση στην συνετή σας κρίση και με βάση αυτά που είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είπε ότι έχουμε να κάνουμε με εκρεμείς ε, πληροφορίες σε σχέση με τα υποπροστασία ε, ήδη υπάρχει διαδικασία αναστολής, δικαστικής αναστολής και νομίζω ότι δεν πρέπει να κλείσει η αναφορά. Εάν θέλετε όμως να κλείσει, τότε θα ήθελα οι ετούντες, οι αναφέροντες να υποβάλουν άλλη αναφορά που να αναφέρεται στο σκέλος που δεν έχει απαντηθεί. Yeah. Ε, ναι. Μιλάμε εδώ για νέα αναφορά ήδη. Είτε πρόκειται εκεί αυτή ή κάποιοι άλλοι που θα την καταθέσουν. Βεβαίω, ο καθένας μπορεί να καταθέσει αυτό που θέλει, αλλά θα είναι μια νέα αναφορά, μια άλλη αναφορά η οποία θα αναφέρεται μόνο σε αυτά τα οποία είπε η Επιτροπή. Τώρα απευθύνομαι στις τέσσερις ομάδες. Δεν μπορώ να μιλήσω εκ μέρου τη κυρία Σαγιαλά. Η ομάδα των σοσιαλιστών θα πρέπει επίσης να λάβει θέση ως προς το θέμα αυτό. βεβαίω. Ναι, ναι, ναι, θα λάβετε τον λόγο κύριο Ματώ, η κυρία Γκρουνή. Είναι σαν αγιά. Έχω απλώς μια παρατήρηση να κάνω σε σχέση με τα όσα είπατε ω πρόεδρο ή ω μέλο. Ε, βεβαίως υπάρχουν δύο ξεχωριστά θέματα, αλλά εδώ μιλάμε για κάτι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στην αναφορά. Ω προ την ανάλυση θα πρέπει να κλείσουμε την αναφορά αυτή, η οποία ε, ενδιαφέρει ένα θέμα που δεν μας αφορά πλέον. Ε, πρόκειται για μια διοικητική διαδικασία που η Επιτροπή θα πρέπει να διευκρινίσει με τον ένα ή άλλο τρόπο και ταυτόχρονα η δική μας Επιτροπή δεν πρέπει να συνεχίσει με αυτή την αναφορά. Όσον αφορά τώρα στην νομοθεσία για τα προστατευόμενα ήδη, αυτό είναι κάτι το ξεχωριστό εφόσον πρόκειται για ένα φάκελο με τον οποίο ασχολούμεθα εδώ και πέντε χρόνια και όταν ένα πρόβλημα διευθετείται ένα άλλο παρουσιάζεται εφόσον αυτό το πρόγραμμα δεν ε, προχωράει για διάφορους λόγους ε, οι πολίτες των ε, Καναρίων που εδώ εκπροσωπούνται είπαν διαμέσου του Κοινοβουλίου ότι υποστηρίζουν το πρόγραμμα αυτό. Υπάρχει μια συμφωνία, υπάρχει μια εξήγηση νομιθετική ε, που ψηφίστηκε από το νόμιμο όργανο, το Κοινοβούλιο των Καναρίων Νήσων, που διευθέτησε τα προβλήματα σχετικά με τα προστατευόμενα είδη που υπάρχουν στην περιοχή. Βέβαια, μπορούμε να αμφισβητήσουμε αυτή την απόφαση, αλλά ήταν απόφαση του Κοινοβουλίου των Καναρίων Νήσων και μετά τα δικαστικά όργανα και τα νομοθετικά υπάρχουν ακριβώς για να ρυθμίσουν το πρόβλημα. Νομίζω ότι η Επιτροπή Αναφορών θα έπρεπε με κοινό νου να κλείσει αυτή την αναφορά. Αλλά βεβαίως κάθε πολιτική ομάδα μπορεί να σκεφτεί να ξανανοίξει αυτή την αναφορά ή να συνεχίσει με μια άλλη αλλά αυτή η αναφορά για την αναξαρτησία του παρατηρητήριου είναι κάτι άλλο. Αυτό το παρατηρητήριο είναι κάτι ε, το ανεξάρτητο και βεβαίως θα μπορούμε, όπως είπαν άλλοι συνάδελφοι, να ξανανοίξουμε αυτήν ε, την αναφορά ή να ανοίξουμε μια αναφορά για άλλα θέματα και να κλείσουμε αυτήν. Ευχαριστώ. Εφόσον ε, δίνω τον λόγο στην κυρία Άγιολα, θα έχουμε μια μακρά συζήτηση. Η κυρία Γκρινή ίσως. Ναι, θα ήθελα να εκφράσω την υποστήριξή μου εξ ονόματος της ομάδας μου. Ζητάω να κλείσει αυτή η αναφορά ε, και για λόγους διαφάνειας πρόκειται για μια... Όχι, κυρία Οκάν, όχι. Όταν θα πάρετε το λόγο θα μιλήσετε. Αλλά όχι, όχι, δεν είναι. Είναι κακόχουστο αυτό το οποίο κάνετε. Με συγχωρείτε που σας το λέω. Μπορεί να έχετε μια γνώμη, δικαίωμά σας, αλλά δεν μπορείτε να έχετε γνώμη για τη δική μου χώρα. Αυτή, αυτό είναι πολύ κακόχουστο. Είχαμε ήδη αυτή τη συζήτηση. Δέχομαι τις... Ε, τα όσα είπατε. Συνεχίζω. Πάντως πιστεύουμε ότι αυτή η αναφορά δεν είναι αναγκαία, μπορεί να υπάρξουν άλλες με περιεχόμενο που θα είναι ίσως διαφορετικό. Και θα ήθελα επίσης να σας ζητήσω, εάν υπάρχουν αναφορές, θα μπορούμε να εργαστούμε μαζί, από κοινού και προσωπικά. Δεν πιστεύω ότι πρέπει να περάσουμε σε ψηφοφορία. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητη η ψηφοφορία. αν πρέπει να υποστηρίξουμε μια πολιτική δράση, μπορούμε να έχουμε τέτοιου είδους συζήτηση. Αλλά πιστεύω ότι τα έχω ήδη πει αυτά στο παρελθόν. Ευχαριστώ η κυρία Γκρινή, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ επιβεβαιώνω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτή την αναφορά διότι η απάντηση δόθηκε μετά για τα προβλήματα τα περιβαλλοντικά που αναφέρεται όντως είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς μπορούμε να παρακολουθήσουμε αλλά στα πλαίσια μιας άλλης αναφοράς εδώ ειλικρινά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε η ψηφοφορία δεν είναι αναγκαία, αλλά έχουμε πάντοτε μια άτυπη ψηφοφορία ζητώντας τη γνώμη του καθενός και μετά ο πρόεδρος βλέπει ποιο είναι το αποτέλεσμα. Ε, κυρία Ευχαριστώ ε, κύριε Πρόεδρε. Εφόσον βλέπω ότι αναφέρθηκε ψηφοφορία προηγουμένως, θα, θα ήθελα να πω κάτι σε σχέση με την προηγούμενη ψηφοφορία. Νομίζω ότι είναι λογική η πρόταση σας να κλείσουμε αυτή την αναφορά και αν υπάρξουν άλλες αναφορές να τις αναλύσουμε και να συνεχίσουμε με τις άλλες αναφορές. Υπάρχει κάτι το οποίο δεν καταλαβαίνω γιατί δεν είχαμε την ίδια διαδικασία για την προηγούμενη αναφορά όταν ο κύριος Στογκαής έκανε παρόμοια πρόταση για να αποφύγουμε την ε, ψηφοφορία η οποία απογοήτευσε πολλούς από τους συναδέλφους μας και τους έδιωξε. Δίνω το λόγο στους αναφέροντες. Λυπάμαι που όλοι διαβάζουν απ' έξω το μάθημά τους και στην πραγματικότητα κανένας δεν μας ακούει δεν άκουσε κανείς τον αναφέροντα. Θα επαναλάβω, γιατί νομίζω ότι δεν έγινε απόλυτα κατανοητό αυτό που είπα. Το περιβαλλοντικό ίδρυμα de Γραναντίγια θα πρέπει να ε, εποπτεύει τα αντισταθμιστικά μέτρα της Κομισιόν. Υπάρχει ένα διορθατικό ε, μέτρο που είναι το Bypass the Arena, όπου όχι μόνο δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα, αλλά όπως ελέγχθη αυτό το έργο δεν θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί και ποτέ αυτό το παρατηρητηρίο δεν είπε ότι ε, αυτό το διορθωτικό μέτρο δεν θα λάβει χώρα. Ποτέ δεν μας το είπε. Ποτέ το Ίδρυμα και εγώ σέβομαι τον κύριο Μάτο, αλλά ε, ελέγχθη ότι το Ίδρυμα υποστηρίζει την ε, κυβέρνηση των Καναρίων νήσων. Εμείς είπαμε και είπατε ότι εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ανεξάρτητο Ίδρυμα. Αυτή η υποστήριξη όμως αμφισβητήθηκε από το Ανώτατο Συνταγματικό ε, Δικαστήριο των Καναρίων νήσων ιδιαίτερα ως προς την απομάκρυνση από τον κατάλογο εκατοντάδων υποπροστασία ειδών που προϋπήρχαν στον κατάλογο. Υπήρχαν ε, και πολλά άλλα ζητήματα και εγώ ήμουνα εδώ όταν εσείς κύριε Μάτο είχατε έρθει ως πρόεδρος του Κοινοβουλίου των Καναρίων Ίσων και είχαν προσέλθει και πολλοί άλλοι πολιτικοί τότε. Και πολλοί σήμερα είναι υπόδικοι για διαφθορά. Μιλήσαμε και για την υπόθεση της Γκρανταρίγια. Μπορούμε να μιλήσουμε και για τα προβλήματα του κύριου Εστρενόρ που ήταν ε, ε, ο διοικητής των λιμενικών αρχών της Γκραναντίγια. Αυτό συμβαίνει γύρω από το που έρτονται Γκραναντίγια. Δυστυχώς. Και φοβούμεθα ότι το ίδιο θα γίνει και με το Ίδρυμα και το Παρατηρητήριο γιατί δεν λέω ότι υπάρχει άμεση διαφθορά, αλλά υπάρχει πολιτική επιρροή, γιατί δεν τιμάται το πνεύμα του Ιδρύματος, το οποίο είναι ένας ανεξάρτητος οργανισμός που εποπτεύει το έργο. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, λέει ο Προεδρεύων. Σας παρακαλώ ησυχία. Εν πλήρη ηρεμία. Αλλά θα ήθελα να σας πω ότι απορρίπτω και θεωρώ ε, λυπηρό ότι ο αναφέρον δεν αναφέρεται στο πολιτικό μου κόμμα, ούτε στη Σάντα Κρούς ούτε στο Πουέρτο Ντεγκραναντίγια. Κανένας δεν είναι υπόδικος από το δικό μου πολιτικό κόμμα. Κανένας ε, δεν κατηγορείται για διαφθορά. Και θα αποφασίσουν τα δικαστήρια. Αλλά εάν δεν σεβόμαστε τα δικαστήρια, για όσα έχουμε επιτάπητος, τι να πω. Όχι, δεν είπαμε απ' έξω το μαθήματάκι μας όπως μας κατηγορείτε. Είπαμε ότι το Ίδρυμα είναι ανεξάρτητο, δεν είναι ανεξάρτητο, υποστηρίζεται από την κυβέρνηση. Εμείς είπαμε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο είπε το ακριβώς αντίθετο. Δηλαδή αποφάσισε και, θεώρησε ότι το Ίδρυμα δεν είναι ανεξάρτητο. Αυτό τουλάχιστον μας λέτε. Το Ίδρυμα λέει αυτά που πρέπει να πει, όπως λένε και οι περιβαλλοντολόγοι. Και να μην αρέσει στον αναφέροντα, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις νομιμοποίησαν ένα όργανο το οποίο ε, λειτουργεί νόμιμα και εργάζεται έτσι ώστε να βγαίνουν καλά αποτελέσματα. Δεν είπαμε το μαθηματάκι μας απ' έξω, προβάλλουμε απ' τα επιχειρήματα. Νομίζω ότι συζητήσαμε παρκώς το ζήτημα. Θέλετε να ψηφίσουμε. Εάν θεωρείτε ότι κλείνει η αναφορά, τότε ε, δυνάμει της παρέμβασης επιτροπής μπορείτε να υποβάλλετε άλλη αναφορά με βάση τα νέα δεδομένα, έτσι ώστε να αποφύγουμε την ψηφοφορία. Γιατί πλησιάζουν και Χριστούγεννα, ε? μην ξεχνάτε. Αυτό το κάνετε προσωπικά ή ως πρόεδρος της Επιτροπής. Κύριε Μάτο, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, όταν προεδρεύει κάποιος, εκφράζει άποψη ως προεδρεύων. Είναι αυτονόητο. Είναι αυτονόητο. Ναι, επειδή το είπατε και πριν, όταν δεν προεδρεύατε. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να επικαλεστώ τον ε, κανονισμό. Μιλώ ως ε, προεδρεύων. Ευχαριστώ τους αναφέροντες και θα ήθελα να τους ζητήσω να επαναπροσδιορίσουν την αναφορά, να την επαναδιατυπώσουν. Κύριε Μάτο, ζητάτε το λόγο, παίρνετε το λόγο χωρίς να στον έχω δώσει, θα σας τον έδινα όμως, με μεγάλη χαρά. Επιμένω όμως ως προεδρεύων ότι θεωρούμε ότι κλείνει η αναφορά και ζητούμε από τους αναφέροντες να επαναδιατυπώσουν μία αναφορά ε, μετά από τις υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σας ευχαριστώ.